Eh. Καλησπέρα συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε την συνεδρίαση, την απογευματινή της Επιτροπής μας και θα ξεκινήσουμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης που αφορά την εφαρμογή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του εμπορίων ανθρωπίνων όντων και προστασία των θυμάτων των έμφυλων αυτών αδικημάτων. Η κυρία Μπερντέρ είναι η συγγήτρια. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Έχετε το λόγο λοιπόν, η συγγήτριά μας, κυρία Μπερντέρ. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα και σας άφησα να περιμένετε. Καλώς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να σας δώσω μια περιγραφή του σχεδίου έκθεσης και θέλω να ευχαριστήσω την, ε, την Άντζελα της Γραμματείας και τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου και τους συνάδελφους στην, Ευρωπαϊκή, στην Υπηρεσία Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την EPRS. Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες βλέπετε και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των εμπειρογνωμόνων που ετοίμασαν την έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο μπόρεσε να ετοιμάσει αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η πρόοδος της οδηγίας και ε, ποια θα είναι η στρατηγική μετά το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε για κάποιες ενδιαφέρουσες εκθέσεις που αναμένονται τον επόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποχρεούνται να εκπονήσει σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας καθώς και συμπληρωματικέ ειδικέ μελέτες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον από τη δική μας οπτική γωνία είναι η μελέτη για την έμφυλη διάσταση του εμπορίου ανθρώπων, όπου εκεί μια σύνοψη έχει διατεθεί και με πλήρης έκθεση θα διατεθεί σύντομα. Ως εισηγήτρια είχα πρόσβαση στην αλογοέκθεση πριν ολοκληρωθεί επισήμω και κατάφερα να συμπεριλάβω κάποιε από τις προτάσεις της εκθέσεως στη δική μας αξιολόγηση για την οδηγία. Η οδηγία εν γέννη είναι πολύ καλό νομοθέτημα. Επικεντρώνεται επί των θυμάτων και επί των βιοπραγιών βάσει το φύλλο. Όμω υπάρχει κενό μεταξύ προθέσεω οδηγία και τη εκτελέσεω τη οδηγία σε προβάσκα των μελών. Η επιτόπια κατάσταση χρήζει βελτιώσεων για να ευθυγραμμιστεί η κατάσταση με τους όρους της οδηγίας. Μέχρι τώρα όλα τα κράτη-μέλη που δεσμεύουν την οδηγία πέρα από τη Γερμανία, εκτό Γερμανία, κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενσωμάτωσαν την οδηγία στην Εθνική Ανομή Τάξη. Προσπάθησα να εστιαστώ επί του συγκεκριμένου θέματο και να κάνω διακρίσει μεταξύ διαφόρων ζητημάτων που όμω επικαλύπτονται. Οι μετανάστε είναι πιο ευάλωτοι στο εμπόριο των ανθρωπίνων όντων, των ανθρώπων κυρίως ε, άνθρωποι χωρίς ε, ε, ταξιδιωτικά έγγραφα και υπάρχει νομική διάκριση όμως μεταξύ εμπορίου ανθρώπων και ανθρωπίνου λανθρεμπορίου. Η συνένεση είναι το βασικό θέμα και που δεν είναι δυνατόν να δώσει κανείς συνένεση ούτως ώστε να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου. Αυτό που να το έχουμε υπόψη μας. Βασικά στιάζεται η έκθεση επί της εμπειρίας των θυμάτων του εμπορίου ανθρώπων. Ακριβή στατιστικά στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν, όπως γενικά για το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά η έκθεση του κ. Στατου 2015 διαπίστωσε το 2010 και μέχρι το 2012 30.146 30.146 θύματα κατεγράφησαν από τα κράτη-μέλη. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων βεβαίως θα είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι συμπεριλαμβάνονται τα θύματα εκείνα που ποτέ δεν εντοπίστηκαν, δεν ταυτοποιήθηκαν. Δεν θα σε εκπλήσει το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν σημαντική έμφυλη διάσταση στο εμπόριο ανθρώπων. 80% των κατοχωρηθέντων θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια. Σαφές παράδειγμα της βίας κατά των γυναικών, λοιπόν. Και εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος ορισμός και εφαρμογή της προσέγγισης που ακολουθεί ε, τη ρήμη ευαισθησία του φύλου. Ζητήσαμε να δώσει κατευθυντής γραμμές περιβαλλτής των πρακτικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύξουμε εμπειρία όσον αφορά την διάσταση του φύλου στην επιβολή του νόμου. Και θέλω να συνεργαστούν τα κάτι μέλη του Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταρτήσουν εκείνους που έρχονται σε επαφή με τα θύματα και να είναι ευαίσθητοι όσον αφορά τα εγκλήματα που διαπράττονται με βάση το φύλο. Συμπεριέλαβα τέτοιους επαγγελματίες για να δείξω που είναι τα κενά. Ο κατάλογος επουδενή δεν είναι όμως εξαντλητικός και αποκλειστικός. Πολλά κράτη-μέλη φαίνεται να παλεύουν με την ιδέα ε, των υπηρεσιών που απευθύνονται στο συγκεκριμένο φύλλο. Διότι δεν είναι σαφές τι εννοούμε με αυτό. Η οδηγία αυτή καθ' αυτή σημειώνει τα θύματα διαφορετικών φύλων, από το αντικείμενο εμπορίου διαφορετικού σκοπού και ποικιλοτρόπω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε την έμφυλη διάσταση του εμπορίου ανθρώπων και βρήκε ότι οι βλάβε που συνδέονται με διάφορε μορφέ εμπορίου είναι διαφορετικέ και η προσέγγιση όσον αφορά τα θύματα θα πρέπει να ταιριάζει ανάλογα. Τα διάφορα είδη λοιπόν του εμπορίου λαμβάνουν χώρα ανάλογα με την προσωπικότητα των θυμάτων και είναι η έμφυλη διάσταση που είναι σαφής. Οι γυναίκε και τα κορίτσια αποτελούν το 95% όλων των θυμάτων του εμπορίου για σκοπού σεξουαλική εκμεταλλεύσεω. Και η μελέτη συμπεραίνει ότι οι βλάβε που συνδέονται με αυτού του είδου το εμπόριο είναι μεγαλύτερε Συνεπώς αυτά τα θύματα θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης ε, βοηθεία. Η οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και να παρέχεται έγκαιρα βοήθεια και στήριξη. Όλα τα κράτη-μέλη φαίνεται να έχουν μηχανισμούς επισήμους που έχουν δημιουργηθεί. Αλλά η επιτόπια κατάσταση ποικίλει και κατά πολύ θα εκπίσει κανέναν αυτό. Ε, ταυτοποίηση των θυμάτων είναι ο πιο προβληματικός τομέας εφαρμογής της οδηγίας και πάρα πολλά θύματα εξακολουθούν να ξεφεύγουν από το δίχτυ καμιά φορά για πολιτικούς λόγους όπως σημειώνεται στην έκθεση πάρα πολλές φυλακές και κέντρα κρατήσεως τελικά δεν δίνουν καλές πληροφορίες για, τα, για τους έγκλειστους εκεί. Ε, λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί επανειλημμένα είναι ότι τα θύματα του ανθρωπίνου εμπορίου έχουν, δικαιώμα, ε, έχουν κάποια δικαιώματα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να προστατεύονται αυτά ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής στη χώρα προέλευσης ή αδίποτε συμπληρωματική διάκριση. Το να μην εντοπιστούν, ταυτοποιηθούν τα θύματα εν πρώτης, αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο στις προσπάθειες αντιμετωπίσεως του εμπορίου ανθρώπων. Για να διευκολύνουμε τον εντοπισμό των θυμάτων θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση και σχετικές πρωτοβουλίες, καλύτερη κατάρτιση για όλο το αρμόδιο προσωπικό, κυρίως εκείνους όπου έχουν προβλήματα, έλλειψη γνώσεων σε αυτή τη φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει εκπονήσει διάφορα έγγραφα, ούτω ώστε να δώσει συμβουλές για την ε, καλύτερη ενίσχυση και βοήθεια για τα θύματα αυτά των εμπορίων ανθρώπων. Ζητούμε να λάβουν υπόψη τις ευρύτερες εξελίξεις και να διαδώσουν τέτοια, να διαβιβάσουν τέτοια έγγραφα, να μοιράσουν. Επίσης τονίζουμε ότι η χρηματοδότηση για ομάδες που εργάζονται και βοηθούν τα θύματα ανθρωπίνου ε, εμπορίου θα πρέπει να δίδονται σύμφωνα με την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και όχι επιβάσεω ιδεολογική. Με τόσε πολλέ οργανώσει, κυρίω οι οργανώσει γυναικών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να είναι ει βάρο των δράσεων για τα θύματα του εμπορίου ανθρώπων. Τα είδη των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν προς τα θύματα περιγράφονται στην οδηγία. Όμως, για μία ακόμη φορά στην πράξη, υπάρχει τεράστια διαφορά από χώρα σε χώρα, όπως και η μέθοδος ε, παροχής των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες επίσης ποικίλουν πολύ όσον αφορά τα είδη του εμπορίου και το φύλλο των εμπλεκομένων ανθρώπων, δείχνοντα στοιχεία ότι τα σενικά θύματα του εμπορίου ανθρώπων ε, είναι πιο δύσκολο να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες όπως στέγαση και εξειδικευμένες υπηρεσίες για φιλομεταβατικά θύματα φαίνεται να μην υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκε και κορίτσια. Θα πρέπει να παρέχονται όμω για όλα τα θύματα επαρκή υπηρεσίες ανεξαρτήτω φύλου. Από τη στιγμή που εντοπιστούν τα θύματα θα πρέπει συστηματικά να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα περίοδου προβληματισμού και ανακάμψεως που δεν είναι αρκετά μεγάλη σε διάρκεια στα κράτη-μέλη, κυρίως για θύματα σεξουαλικής εκμεταλλεύσεως με μεγαλύτερες βλάβες. Βεβαίω δεν πρέπει να λησμονούμε ότι βασικό πυλώνα είναι η πρόληψη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση για τι υπηρεσίε των, θεμα... θυμάτων του εμπορίου ανθρώπων. Χρειάζονται εξαρτήσει ευαισθητοποίηση που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικέ εάν έχουν συγκεκριμένου στόχου αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να γίνουν εκστρατείε για να ευαισθητοποιηθεί ευρύτερο το το κοινό για να γίνονται σωστές ηθικές ε, επιλογές. Δεν αρκεί όμως, θα πρέπει να υπάρχει σωστή κατανόηση της ζήτησης, ούτως ώστε τελικά να φτάσουμε στην καρδιά του προβλήματος και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτό όλος ιδιαίτερος εστιαζόμενοι επί του εμπορίου παιδιών και να εκδώσει προσανατολισμούς ευαισθήτους όσον αφορά το φύλλο, βάσει το άρθρο 18.4 της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την ποινικοποίηση της χρήσεως την γνώση των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των θυμάτων των εμπορίων ανθρώπων. Οι υπηρεσίε που είναι άμεσο αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεω θα πρέπει να ποινικοποιηθούν. Όμω ίσω δημιουργούνται νομικά προβλήματα για την απόδειξη της γνώσεως του χρηστου καποια Κάποια κράτη-μέλη έχουν κινηθεί από αυτού Κάποια άλλα κρατημέλη έχουν εμείς μείνει πίσω. Συνάμει τι οδηγίε ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει εκθέσει από αυτό. Θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένε δράσει από αυτή τη βάση των πολισμάτων σχετικά με τι διάφορε δράσει και να δει πώ οι δράσει επηρέασαν τη ζήτηση για τι υπηρεσίε που παρέχονται τα θύματα των εμπορίου ανθρώπων. Όπω πάντα, ζητώ λεπτομερέστερα στοιχεία, συνεπιστοιχεία, για να διαμορφώσουν πολιτικέ βάσει στοιχείων. Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να παρέχουν στοιχεία κατά υποκατηγορίε, άλλα κράτη-μέλη όμω παρέχουν τα ελάχιστα στοιχεία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε όλα αυτά, ζητώντα από όλα τα κράτη-μέλη να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία, τα οποία θα είναι κατά ηλικία, φύλλο, είδο εκμετάλλευση χώρες προελεύσεως και προορισμού. Μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα. Θα πρέπει επίσης να συλλέγουμε στοιχεία όσον την πρόσβαση στα δικαιώματα και τις υπηρεσίες για τα θύματα. Και εθνικοί εισηγητέ που έχουν, έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω οδηγίας έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν όσον αφορά τη συλλογή των πληροφοριών. Βεβαίως, η φύση της εκθέσεως σημαίνει ότι περιοριζόμαστε όσον αφορά αυτά που μπορούμε να πούμε, όπως πάντα, και κάποια στοιχεία λοιπόν έχουν καλυφθεί εντάχει για να περιορίσουμε το μήκος του κειμένου. Προσβλέπω στις τοπολογίες και προβλέπω σε σημαντική συζήτηση μαζί στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπέρντερ. Ξεκινάμε με το γύρο παρεμβάσεων από τους κοιόδης εισηγήτες. Εξ ονόματος του ΕΛ και η κυρία Κοράτσα Μπέρντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ Κάθριν Υποστηρίζω πάρα πολύ την προοπτική της ενσωμάτωσης της ε, ισότητας των φύλων σε αυτή την έκθεση, γιατί η πλειοψηφία των θυμάτων ανθρωποεμπορίας είναι τα κορίτσια και οι γυναίκες. Δράτω με τις ευκαιρίες να αποτίσω φόρο τιμής ε, στον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου λαθροεμπορίας ανθρώπων, επικεντρωνόμενη στις γυναίκες ε, και στα παιδιά. Πρέπει να εστιαστούμε στην υλοποίηση, στην εφαρμογή, να αξιολογήσουμε αν εγκληματοποιούν, ποινικοποιούν επαρκώς την λαθρεμπορία ανθρώπων ή ε, τα κράτη-μέλη ή αν δημιουργείται ένας πολιτισμός ε, χαλαρότητας και ατιμορρησίας. Πρέπει να εστιαστούμε και στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της ανθρωποεμπορίας και την προστασία επίσης των θυμάτων. Δυστυχώς υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ όλων της αυξανόμενης ανθρωποεμπορίας και των, της μετανάστευσης. Πρέπει να δούμε την κατάσταση των γυναικών. Κανείς δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, ή κακομεταχείρισης. Ε, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Είναι ιδιαίτερα δραματική η κατάσταση για τα παιδιά. Η Ευρωπόλ πρόσφατα ανέφερε 10.000 παιδιά πάνω κάτω. Είναι τρομακτικός αυτός ο αριθμός, φρικτός εξαφανίζονται 10.000 παιδιά όταν εισέρχονται στην Ευρώπη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πορνείας, κακομεταχείρισης. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η καταχώρηση, η καταγραφή παιδιών ε, είναι ένας τρόπος να ενταχθούν σε ένα σύστημα προστασίας. Και έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να διατηρούμε τα ίχνη τους, να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να εντοπίσουμε που βρίσκονται. Είναι η ανθρωπεμπορία ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και απαιτεί συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Χρειάζονται όλα τα μέσα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Κάποια κράτη-μέλη κάνουν αρκετά για τη συνεργασία αυτή, η συνεργασία αστυνομική, δικαστική με την Ευρωπόλ, Eurojust, Frontex και φυσικά με το συντονιστή κατά του ανθρωποεμπορίου. Κάνουμε αρκετή χρήση των hotspots για τον εντοπισμό γυναικών που θα μπορούσαν να είναι ευάλωτοι στόχοι ώστε να τις εκμεταλλεύονται αυτοί οι ε, έμποροι ανθρώπων. Και πρέπει εδώ να δούμε ότι πρέπει να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καταπολεμήσουμε αυτούς τους ε, ανθρωποεμπόρους. Και όπως αναφέρθηκε η συλλογή στοιχείων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι ένας τρόπος να εντοπίσουμε πιθανά ενδυνάμει θύματα και να προλάβουμε εγκλήματα. Επίσης ε, πρέπει να αυξηθεί η δράση μας ε, Υπάρχει σαφώς πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Πρέπει να δοθούν περισσότερα εργαλεία και εργαζόμαστε ως Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό για να έχουν μέσα και εργαλεία στα χέρια τους να υπάρξει η δημιουργία αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης και ανταλλαγής πληροφοριών. Η Κάθριν ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και υπαλλήλων, διοκτικών αρχών και άλλων που πρέπει να συνδράμουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους μετανάστες, τα κορίτσια, θύματα δηλαδή ανθρωποεμπορίου, στην πρόληψη κιόλα, ε, στη φάση της πρόληψης. Πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με το ζωφερό, το σκοτεινό διαδίκτυο, τι μπορούμε να κάνουμε με νέες τεχνολογίες ε, για να εντοπίσουμε, ανοιχνεύσουμε και καταπολεμήσουμε, ακόμα και να προλάβουμε τέτοιου είδους κατάχρηση του διαδικτύου σε, ε, με όσους εμπλέκονται σε αυτό, με τα μέσα και εργαλεία που θα εκπονήσουμε. Είναι σημαντικό να δούμε αν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα νομικά μέσα όσον αφορά την αναγνώριση αμοιβαία δικαστικών αποφάσεων και νομολογίας εντολών προστασίας ε, για τις γυναίκες, ε, εντάλματα σύλληψης, ε, εντολή ανακριτική για την Ευρώπη, ευρωπαϊκή ανακριτική εντολή. Το θέμα δηλαδή της κατάσχεσης επίσης των περιουσιακών στοιχείων των ανθρωποεμπόρων και οι ποινές και κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται. Έχουμε εδώ τεράστια ποσά, 150 δις δολάρια ετήσια εις βάρος ουσιαστικά των γυναικών και των κοριτσιών ε, στις πλήστες των περιπτώσεων. Θα είναι σημαντικό να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε διακομματικά, υπερκομματικά, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η τρομερή μάστιγα και τα κράτη-μέλη επιτέλους, γιατί για τα κράτη-μέλη πρόκειται να υπομισθούν τις ευθύνες τους, να εφαρμόσουν όλες τις πτυχές της οδηγίας για την καταπολέμηση του ανθρωποεμπορίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία Κοράτσα. Ελπίζω ότι η πτήση σας θα φύγει στην ώρα της και θα έχετε και καλό ταξίδι όπως σας εύχομαι. Τώρα η κυρία Χόνιμπολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την εξαιρετική της ε, ε, έκθεση. Έγινε μία στο θέμα της ε, συνεργασίας και έχω την αίσθηση ότι η έκθεση αυτή συνιστά μια πολύ καλή βάση για συνεργασία και θα συνεργαστούμε τις άλλες πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό. Το έχουμε ήδη κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον, γιατί είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Γιατί όπως υπόθηκε θα πρέπει όλες οι χώρες μέλη να συμμετάσχουν ενεργά, περισσότερο από ό,τι το έχουν πράξει στο παρελθόν, ούτε ώστε να έχουμε μικτές ομάδες. Δυστυχώς η Επιτροπή καθυστέρησε με την έξεση εφαρμογής, αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα σημεία σύντομα και ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε και εμείς να συμπεριλάβουμε τα δικά μας ε, σημεία ε, με την υποστήριξη των συντονιστών κατά του τράφικινγκ. Μιλήσαμε για μια αποτελεσματική ταυτοποίηση των θυμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για θύματα και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις γιατί πολλά από αυτά τα θύματα απλούστατα δεν εμφανίζονται, δεν μπορούν να ανεβρεθούν και να ταυτοποιηθούν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερες διαδικασίες, γιατί αυτό θα είναι κλειδί για τη μείωση της εμπορίας ανθρώπων. Και τα ίδια τα θύματα χρειάζονται κάτι τέτοιο. Μιλάμε για γυναίκες ιδιαίτερως, αλλά πρόκειται και για γυναίκες και κορίτσια, τα οποία γίνονται αντικείμενο εμπορίας ε, σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν Διαφορετικέ ανάγκε. και όλο αυτό το στοιχείο θα πρέπει να συμπεριληφθούμε στη διαδικασία ταυτοποίηση. Ε, τα θέματα είναι πολύ σημαντικά σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο επειδή είναι σήματα και επειδή έχουν διάφορες και σημαντικές ανάγκες, επειδή μπορούν επίσης να εισφέρουν, να συμβάλλουν στην πρόληψη, στην ε, αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ περισσότερο τι γίνεται με τα θύματα και να μην τα αντιμετωπίσουμε απλώς και μόνο θύματα, αλλά σαν ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν εξαιρετικά στην προσπάθεια πάταξης του, αυτού του φαινομένου. Αυτό έχει καθοριστική σημασία, γιατί οι έμποροι ανθρώπων, οι διακινητές, είναι οργανωμένοι εγκληματίες. συμμετέχουν στο οργανωμένο έγκλημα, άρα λοιπόν εκμεταλλεύονται τα πάντα ούτως ώστε να ε, υλοποιήσουν τις εγκληματικές τους ε, προθέσεις. Κάνουν χρήση και του διαδικτύου. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν και εκείνοι και να τους ανοιχνεύσουμε μέσω αυτών των δικτύων οι αστυνομικέ δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συντονιστούν και να προσαρμοστούν στα μέσα και τα εργαλεία που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες. Δεν θα πρέπει μόνο να συμμετάσχουν οι χώρες μέλη και οι κυβερνήσεις, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι επίσης τα όργανα εφαρμογής του δικαίου ε, πραγματικά ε, είναι προσελωμένοι στο στόχο μείωσης της εμπορίας ανθρώπων. Γιατί έχει μεγάλη σημασία κάτι τέτοιο, γιατί προφανώς οι διακινητές θα πρέπει να αναγνωριστούν, θα πρέπει να εντοπιστούν και να θεωρηθούν ως εγκληματίες. Είναι ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα αυτή η πράξη. Το άρθρο 33 αφορά την ε, ποινικοποίηση όσων ε, ε, χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες. Και θα πρέπει πραγματικά να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να θεωρηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη εγκληματική και αξιόπινη πράξη εμπορία ανθρώπων η έκθεση αυτή καθ' αυτή επικρίνει το γεγονός ότι η χρήση των υπηρεσιών εμπορίας ανθρώπων δεν συνιστά μέχρι στιγμής ε, ξεκάθαρα μια ε, αξιόπινη πράξη. Τα νούμερα πραγματικά όσον αφορά το τράφινγκ είναι φρικιαστικά. Ε, η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ο βασικός στόχος ε, αυτό συνεχίζουμε να το λέμε γιατί η εμπορία ανθρώπων αφορά πάρα πολύ την εμπορία γυναικών. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, ε, εργασιακή εκμετάλλευση κλπ. Αλλά τα, τα μεγαλύτερα ποσοστά ε, διακινούνται για σεξουαλικούς ε, σκοπούς. 95% από αυτούς είναι γυναίκες. Σχετίζεται λοιπόν πάρα πολύ το θέμα αυτό με, ε, με τη διακίνηση γυναικών με το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 69% των θυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, γυναίκες και κορίτσια και 95% από αυτούς ε, για το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι ο λόγος για το οποίο είναι τόσο σημαντικό εμείς ως ε, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ όλα αυτά τα φαινόμενα και να επακριβήσουμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας και να συνεχίσουμε και το νομοθετικό μας έργο ε, στο πλαίσιο αυτό, ε, ούτως ώστε η βία κατά των γυναικών να θεωρηθεί ξεκάθαρα εγκληματική πράξη. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνεχίσει την εκστρατεία ούτως ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο γιατί η σεξουαλική εκμετάλλευση και η πορνεία συνιστά βία κατά των γυναικών υπό τη μία την άλλη μορφή. Και αυτό με φέρνει στο θέμα της ε, ε, μείωσης της ε, ζήτησης για την εμπορία γυναικών προκειμένου να, ε, προκειμένου να υπάρξει σεξουαλική εκμετάλλευση. γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να εφόσον μειωθεί η ζήτηση γυναικών αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του φαινομένου συνολικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου, να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να αναλάβουμε εδώ έναν ηγετικό ρόλο και, να... και η μείωση της ζήτησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό επιχείρημα. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω την άξη της συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης, την παροχή πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με το θέμα αυτό, γιατί όπως υπόθηκε ήδη η συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με τα θέματα αυτά δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να, να ε, ε, προσπαθούμε εδώ. Γιατί έχουμε την αρχική οδηγία που πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα, είναι εξυγχρονισμένη και περιεκτική και είναι ένα δείγμα αυτού το οποίο μπορεί να επιτευχθεί εφόσον υπάρχει κανοποιητική διασυνοριακή εργασία θα πρέπει να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση και να εξασφαλίσουμε όταν η έκθεση εφαρμογής ε, έρθει από την, ε, φτάσει από την Κομισιόν να πραγματικά να συμπεριλαμβάνει όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία επισημαίνει η δική μας έκθεση. ούτω ώστε να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν με, την, με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει το λόγο η κυρία Λαβιόρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Κάθριν Μπίρντερ για αυτό το έργο που επετέλεσε. Είναι μια εξαιρετική έκδοση αυτή Είμαι και εισηγήτρια για την συντάκτη γνωμοδότηση για την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ. Είναι τερμα, τεράστια σημασία ότι η Επιτροπή μας έχει αρμοδιότητα για το θέμα αυτό και λόγω των στατιστικών στοιχείων που καταδεικνύουν ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες είναι εκείνα που και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης στο μέγιστο βαθμό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικού είδους και διαφορετικοί τύποι ανθρωποεμπορίας και πρέπει να έχουμε διαφορετικές διαφοροποιημένες στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί κάθε τύπος αυτού του φαινομένου. Υπάρχει η καταναγκαστική εργασία, υπάρχει η βιομηχανία του σεξ, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της πορνείας και εκμετάλλευσης ε, εις βάρος των παιδιών. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική ξεχωριστή και για τα παιδιά. Είναι τεράστιο τεράστιας εμβέλεια στο θέμα αυτό και πρέπει η κοινοβουλευτική μας επιτροπή που αντιμετωπίζει, ε, εξετάζει την οδηγία αυτή που υφίσταται και υπό το πρίσμα της ε, ισότητας των φύλων να δραστηριοποιηθούμε και να εξετάσουμε το ανθρωποεμπόριο ενεργά με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτή τη μάστιγα μια και πλήττει με τέτοιο τρόπο γυναίκες και παιδιά και κορίτσια Πρέπει να δούμε λοιπόν μήπως κάποιοι υποστηρίζουν κάποιους εγκληματίες. Οι εγκληματίες ε, πρέπει να διώκονται με την μέθοδο και της πρόληψης. Και όταν κάνουμε λόγο για την πρόληψη πρέπει να υπάρξουν ιδιαίτεροι συντελεστές ε, και εργαλεία. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται, εξωθούνται στο να εκτεθούν γυναίκες και κορίτσια στην ανθρωποεμπορία. Όμως, ε, οι, ας το πω έτσι, έρχονται και ταυτόχρονα εξωθούνται. Υπάρχει εδώ λοιπόν ζήτηση, μεγάλη ζήτηση από πλευράς της βιομηχανίας του σεξ και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ζήτηση για γυναίκες και κορίτσια. Και αυτό εκμεταλλεύονται ακριβώς οι ανθρωποέμποροι, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση αυτών των γυναικών και κοριτσιών. Πρέπει να προχωρήσουμε με βάση την νομοθεσία και να εκπονήσουμε τέτοιου είδους ε, βήματα και διαβήματα ώστε να μπορέσει να καταπολεμηθεί το δίκτυο αυτό, αυτή η μάστεγα, μάστιγα με μέτρα που θα λάβουμε άμεσα τώρα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι απόλυτα κάθετη και ακόμα πιο σαφής ε, ότι αυτό πρέπει να γίνει με κάθε τρόπο. Και φυσικά θα πρέπει επίσης να επιβάλλουμε την ενισχύει νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία. Πρέπει όμως να δράσουμε και με εξειδικευμένο τρόπο αναλαμβάνοντας ε, βήματα και διαβήματα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο εξειδικευμένοι. Και όταν κάνουμε λόγο για ζήτηση, κάνουμε λόγο για άνδρες, για άνδρες που αγοράζουν υπηρεσίες πορνείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και είναι οι πελάτες και τους προσφέρεται το εμπόρευμα εντός εισαγωγικών. Αυτή είναι η φρικτή κατάσταση και έχουμε και ανηλίκους που εμπλέκονται σε όλο αυτό το δίκτυο. Και φυσικά δεν είναι μια ε, κοινωνία ισότητας ή δικαιοσύνης μια τέτοια κοινωνία που έχει τέτοιου είδους ε, καρκινώματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα θύματα και πρέπει να μην υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για αυτή τη δράση μας όσοι είναι θύματα να μην, να μην τιμωρούνται γι' αυτό διότι έχουν εντός εισαγωγικών παραβεί, παραβιάσει νομοθεσία ή διατάξεις όντας για παράδειγμα αν, αν, ε, αν διαμένουν σε μια χώρα και τα λοιπά και ή τις διατάξεις αυτές ίσως τις έχουν παραβεί και πρέπει να δούμε ότι αυτές οι γυναίκες είναι θύματα ανθρωποεμπορίας και είναι όντα θύματα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ειδική τους κατάσταση και να μην τιμωρούνται και από πάνω επιπρόσθετα. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης. Θα έλεγα τούτων λεχθέντων ότι είναι εξαιρετική πραγματικά αυτή η έκθεση και θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια ώστε με κάποιες τροπολογίες να βελτιωθεί και να μπορέσουμε το έργο μας να το προαγάγουμε στην ε, αρμόδια επιτροπή και στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ. Εσείς θέλετε να παρέμβετε. Έχετε τον λόγο λοιπόν κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απλά και μόνο για να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μπέρντερ για το κείμενο. Θεωρώ ότι η έκθεση πολύ καλά εντάσσει πολλές από τις πτυχές που μας ανησυχούν ε, σε σχέση με το θέμα αυτής της οδηγίας. Απλά και μόνο να επιμείνω και να εμείνω σε κάποια σημεία που πρέπει να τονιστούν. Το πρώτο για τη συλλογή των στοιχείων αναφέρθηκε από την εισηγήτρια και είναι σημαντικό. Παρότι έχουμε μια θεσμική δομή για αυτή τη συλλογή δεδομένων και για την διάδοση και διάχυση πληροφοριών. Τουλάχιστον τα δημόσια στοιχεία, τα τελευταία που έχουμε είναι για το 2012. Βρισκόμαστε πολύ πίσω λοιπόν χρονικά, χωλένουμε, ενώ το πρόβλημα είναι μια μάστιγα και το πρόβλημα είναι ένα φαινόμενο που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, περιπλέκεται η κατάσταση λόγω αυτού του ζητήματος. Γενικά έχουμε ένα νομοθετικό μέσο που είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην εφαρμογή και υλοποίηση. Και μεταξύ άλλων πραγμάτων πρέπει εδώ προφανώς ε, και το λέει η έκθεση, τα προβλήματα συντονισμού και τα να δράσουμε αποτελεσματικά. Δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το ότι θα εστιαστούμε στην έκθεση σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν και ίσως απουσιάζουν, έχουμε μια ολόκληρη σειρά φαινομένων που δεν υπήρχαν τότε όταν συντάχθηκε η οδηγία και πρέπει να τα εντοπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Η εκμετάλλευση σεξουαλική κάθε φορά αυξάνεται και είναι όλο και πιο σημαντικό φαινόμενο στους διαδρόμους και διάβλους που ακολουθούν ε, οι μετανάστες. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι θύματα αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει όμως ένα κενό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και να δραστηριοποιηθούμε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το θέμα των ανηλίκων είναι τεράστια σημασία. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ισχυρέ δράσει, αποτελεσματικέ δράσει. Κάποια σημεία επιπλέον όπου με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια που έκανε εξαιρετική δουλειά για να τα καλύψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των ομάδων και θα λάβουν τώρα τον λόγο οι συνάδελφοι, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η κυρία Χέντ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ε, εισηγήτρια. Είναι πολύ καλή η βάση η έκθεσή της ε, για εργασίες. Πολλοί είπαν πολλά καλά πράγματα. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ επί της καταστάσεως. Ήμουν εισηγήτρια για το εμπόριο ανθρώπων το 2011 και τη σχετική νομοθεσία. Και αν συγκρίσει πώς ήταν, με το πώς ήταν η κατάσταση στην αρχή και πώς είναι τώρα, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Δεν ήταν και τότε εύκολη η κατάσταση. Δεν ήταν εύκολο να θεσπίσουμε την κατάλληλη νομοθεσία. Υπήρχαν πολιτισμικά θέματα που δημιουργούσαν προβλήματα. Αλληλουσυγκρούμενες προσεγγίσεις. Δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της πενταετίας προχωρήσαμε πολύ. Και μπορούμε την οδηγία να την αναπτύξουμε έτη περαιτέρω. Χαίρομαι που έχει μπει η ε, διάσταση του φίλου στο κείμενο. Είναι η πρώτη νομοθεσία που έχει μέσα αυτή την πτυχή του φίλου. Αφορά κυρίως γυναίκες και παιδιά. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και στο μέλλον θεσπίσουμε νομοθεσία που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Όχι μόνο όταν μιλάμε για την παιδεία και για την κατάρτιση, αλλά και για άλλα ζητήματα. Τώρα τα παιδιά. Εκεί, σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τα δικαιώματα των παιδιών. Και θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο, διότι ε, βλάπτονται πολύ τα παιδιά, πολλά παιδιά. Εγώ προσπάθησα να δημιουργήσω ένα νομοθετικό κείμενο που θα οδηγούσε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά της αγοράς προϊόντων σεξ. Θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε εκείνους που εν γνώση τους αγοράζουν σεξουαλικής φύσεως υπηρεσίες. Δώσαμε μεγάλη μάχη γι' αυτό. Να γίνει αυτή η αναφορά. Και όπως είπαν και οι Μαλίν και η μέρη, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τη ζήτηση, διότι η ζήτηση είναι το κομβικό σημείο. Και τα περισσότερα θύματα του ανθρωποεμπορίου πρέπει να παρέχουν σεξουαλικής φύσεως υπηρεσίες. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκανδιναβικό μοντέλο που ανέφερε η Μέρη. Θα πολεμήσω γι' αυτό. Όσον αφορά την περίοδο ανάκαμψης, ε, ε, αυτό ήταν και, αυτό και αποκατάστασης και αυτό ήταν ευαίσθητο θέμα. Έγινε μάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το θέμα. Και αυτό θα πρέπει να το προθίσουμε και χαίρομαι που η συγγήτρια το έλαβε αυτό υπόψη σαν στοιχείο. Αναφερθήκαμε σε στατιστικά στοιχεία και θεωρήσαμε ότι τα περισσότερα θύματα ήταν από τρίτες χώρες. Όμως έχουμε εξίσου πολλά θύματα που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να φροντίσουμε να τα καλύψουμε αυτά τα θέματα. Είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά. Εξίσου προβληματική είναι η κατάσταση, είτε θα επιστρέψει το θύμα σε αφρικανική χώρα, είτε θα επιστρέψει στη Ρουμανία. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το, τα μέσα που έχουμε για την ισότητα των φίλων σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να το σκεφτούμε. Το θέτω αυτό στην εισηγήτρια και σε όλους τους άλλους. Εγώ έχω μεγάλες προσδοκίες. Πρέπει να συλλέξουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη Και αυτό κατάφερα να το τονίσω. Δεν τα κατάφερα όσον αφορά αυτό που ήθελα να πετύχω με τη μείωση της ζήτησης. Αλλά κατάφερα να πείσω τα κράτη-μέλη να μας ενημερώσουν για το τι έκαναν, τι προσπάθειες κατέβαλαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο σφιχτή ούτως υπήν η οδηγία, πιο αυστηρή στο μέλλον. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας κάτι. Όταν ξεκινήσαμε την επεξεργασία των θεμάτων αυτών του ανθρωποεμπορίου στη Σουηδία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η αστυνομία στη Στοκχόλμη ετοίμασε μια διάσκεψη για το θέμα. Στείλαν προσκλήσεις σε όλους αστυνομικούς στη χώρα και μέχρι τη Βόρεια Σουηδία, στον Ακτικό κύκλο και ένα αστυνομικό από εκεί έστειλε τρει αστυνομικού στη Στοκχόλμη και ήρθαν από το Βόρειο Πόλο ουσιαστικά από, τον αρχικό κύκλο στη Στοκχόλμη και όταν έφτασαν αυτοί οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ ε, στενοχωρημένοι γιατί ήταν τροχονόμοι για την κυκλοφορία. Traffic police δηλαδή. Που ασχολούνται με το traffic την κυκλοφορία και όχι με το traffic το εμπόριο. Και έγιναν πολλά αστεία με βάση αυτό το λογοπαίγνιο αλλά έμαθαν ε, πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν και εμάς και τους άλλους. Ε, πρέπει να το επεξεργαστούμε αυτό, είναι κάτι που μας προβληματίζει όλους, ε, πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και πρέπει να τολμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να θέσουμε τέρμα στο άνθρωπο εμπόριο και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε αυτό ο γύρο των παρεμβάσεων και τώρα έχει το λόγο εξ ονόματο της Επιτροπής η κυρία Μίρια Βασιλιάδου ε, από, την, ε, από το Γραφείο Συντονισμού για το Τράφικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Καταρχάς καλωσορίζω και την έκθεση και αυτά που καλύπτει η έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος την κυρία Κάθριν Μπέρντερ. Ήταν άριστη η συνεργασία μας. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά ήδη έχουμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ευχαριστώ. Να πω κάποια πράγματα. Καλύφθηκαν κάποια σημεία ήδη στις συνεδρίες Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών χθε το πρωί. Θα εστιαστώ μόνο επί της έμφυλης διαστάσεως του φαινομένου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές, επανειλημμένα το έχουμε αναφέρει ότι το ανθρωποεμπόριο είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα τον έμφυλο και γι' αυτό εντοπίσαμε ότι είναι διαθρωμένη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών το ανθρωποεμπόριο με θύματα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Είμαστε σαφέστατοι, απηχώ λέγοντας το αυτό την άποψη των μελών του Κοινοβουλίου. Για μας το ανθρωποεμπόριο κινείται από δύο παράγοντες. Το χρήμα πολύ ισχυρό παράγων για το οργανωμένο έγκλημα που βγάζει τεράστια κέρδη και, εκείνοι που το, και αυτοί που αναμειγνύονται στους νομικούς κύκλους, ε, νόμιμους κύκλους και για τους παρανόμους. Και μετά η άλλη πτυχή είναι η ζήτηση για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία επί των οποίων εσταζόμεθα. Τους έχουμε δώσει προτεραιότητα. Πριν πω κάτι άλλο, προσέξτε το εξής. Την έκθεση της Ευρωπόλ θα δημοσιευθεί σε μία-δύο μέρες στην ιστοσελίδα της Ευρωπόλ, αν δεν κάνω λάθος. Ήδη έχει μοιραστεί στα κράτη-μέλη. Ό,τι πω από τούδε και στο εξή αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπόλ. Ευχαριστώ τους, το, στη συνάδελφο αναφέρθηκε στην ανάγκη για πρόσφατα στοιχεία. Πράγματι. Η έκθεση της Ευρωπόλ ρίχνει κάποιο φως αυτό αναφέρει διαπιστωθήσεις τάσεις, πολύ πρόσφατες, με στοιχεία του 2015. Για τα στοιχεία λοιπόν συνεχίζεται η προσπάθεια. Συλλέξαμε προκαταπτικά στοιχεία για το 2013. Τα επόμενη συλλογή στοιχείων ξεκινά τώρα. Μεγάλο πρόβλημα η συλλογή στοιχείων. Λόγω θέματος. Κινούμεθα από σωστή κατεύθυνση. Ήδη μπορώ να πω ότι έχουμε ενδείξεις ότι η ποιότητα των στοιχείων έχει βελτιωθεί σε αυτή την φάση που τώρα ξεκίνησε. Για τα παιδιά. Από την οδηγία και από τη στατική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σαφές ότι έχουμε εστιάσει προσπάθειες στα παιδιά. Είναι λυπηρό, κατά την άποψή μου, ότι τώρα, όπως είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, με τα 10.000 αυτά παιδιά Είμαστε, κινούμεθα πολύ αργά στον τομέα των παιδιών. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Τα συστήματα προστασία των παιδιών είναι η σωστή κατεύθυνση για τα κάτι μέλη. Δεν θέλω να χρονοτριβώ. Να σας πω τι κάνουμε τώρα. Σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Τα θέματα της Έχουμε τέσσερα έγγραφα που θα εκδοθούν σύντομα. Το πρώτο. Μελέτη για την έμφυλη διάσταση του εμπορίου. Όπως είπε η κυρία Μπέρντερ. Της διαθέσαμε τη μελέτη. Θα δημοσιευτεί αυτή σύντομα. Ετοιμάστηκε από ένα κονσόρσιουμ πασίγνωστων ακαδημαϊκών, επιφανέστατων ακαδημαϊκών, με μεγάλη εμπειρία, τριακονταετή όσον αφορά αυτού του είδους τη βία. Ελπίζουμε το κείμενο να βοηθήσει. Θα εκδοθεί το κείμενο τον επόμενο μήνα. Έχουμε την έκθεση τάσεων όπως αποκαλείται, ίσως ο τίτλος δεν είναι και τόσο καλός αποτέλεσμα της νομοθεσίας του άρθρου 20. Τα κράτη-μέλη έδωσαν στους συντονιστές τους αρμοδίους τις εκθέσεις τους. Και εμείς συντάσσουμε στο γραφείο μου μια έκθεση που θα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είναι έτοιμη αυτή τις επόμενες εβδομάδες και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με ανακούφιση βλέπω ότι η έκθεση της Ευρωπόλ συνάδει με τα πορίσματά μας. Άρα είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούμε σωστή πορεία. Να τονίσω κάτι. Η κοινωνία των πολιτών εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με την έκθεση. Και η πλατφόρμα για την κοινωνία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συμμετείχε πλήρους εργασίες. Διάφορα κάτι μέλη συμμετείχαν. Οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών συμμετείχαν. Έγιναν πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελήφθησαν δεόντως υπόψη, απόψεις και συμπεριλήφθησαν στην έκθεση. Μετά, η, η έκθεση ε, για την ενσωμάτωση οδηγία της εθνικές ένωμες Τάξης. Ευχαριστώ εκ νέου την Κάθριν Μπέρντερ για τις ερωτήσεις και το ενδιαφέρον της και τις ερωτήσεις που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γραπτή ερώτηση που έλαβε απάντηση. Να σας πω το εξή. Με τη βοήθεια μελέτης συμμόρφωσης που ανετέθη σε εξωτερικό φορέα αναλύουμε τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Η οδηγία είναι πληρέστατη. Ε, βοήθεια, προστασία των θυμάτων, ποινικέ κυρώσεις, πρόληψη, λαμβάνει υπόψη, όλη η διαδικασια διαδικασία είναι δυναμική. Κάποια κράτη-μέλη ολοκληρώνουν την κοινοποίηση. Η Γερμανία ακόμα αναμένεται να δώσει την πλήρη κοινοποίηση για την ενσωμάτωση τη οδηγία στη δική της ανομητάξη. Περιμένουμε τελικά αποτελέσματα τη μελέτη συμμορφώσεω το μήνα Απρίλιο. Πρέπει να αποφύγουμε όμω πολλαπλέ εκθέσει. Χρειάζεται συνέπεια, συνοχή, να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα τη μελέτη συμμορφώσεω. Γι' αυτό η έκθεση για το βαθμό συμμόρφωση των κρατών μελών, άρθρο 23,1 όπω ξέρετε όλοι, θα παρουσιαστεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. Στην έκθεση θα αναφέρονται οι συνέπειες των εθνικών ένωμων τάξεων που θα θεωρεί σαν κολάσιμο, σαν ποινικό αδίκημα την παροχή σεξουαλικών τέτοιων υπηρεσιών. Άρθρο 23, παράγραφος 2. Έχουμε δύο παραγράφους στο νομοθέτημα που καλύπτουν το θέμα. Να πω ότι όσον αφορά την έκθεση ποινικοποίησεως, απηχώ τις απόψεις των, απόψεων των Ευρωβουλευτών δεν συζητούμε τίποτα άλλο παρά την ποινικοποίηση και τις ποινές επιβάλλοντες εκείνου που αναμειγνύονται σε ένα έγκλημα. Όπω το έγκλημα αυτό καθορίζεται, η αξιόπινη πράξη καθορίζεται από τη συνθήκη. Έχουμε και την οδηγία του 2009 για τις κυρώσει επί των εργοδοτών. Εκείνοι που εν γνώση τους χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε επικών τρίτων χωρών που είναι θύματα ανθρωποεμπορίου πρέπει να έχουμε ένα συνεπές νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Αυτά που κάνουμε είναι αρκετά αν δεν επιβάλλουμε ποινικέ κυρώσει σε εκείνους που είναι αμυμένοι στο έγκλημα. Δύσκολο να στοιχειοθετηθούν αυτές οι πράξεις, όπως και σε άλλους τομείς του εγκλήματος. Κάναμε παρόμοιες συζητήσει σε άλλα θέματα, όπως βία κατά των γυναικών, βιασμοί, ε, επιθέσεις σε διαπροσωπικό επίπεδο και 20-30 χρόνια τα κουβεντιάσαμε αυτά. Πώς συλλέγουμε τα στοιχεία. Αυτός δεν είναι λόγος όμως εκείνοι που είναι αναμειγμένοι σε μια αξιόπινη ε, πράξη να μην λογοδοτήσουν και να μην τιμωρηθούν. Τελευταίο στοιχείο. Τι γίνεται μετά το 2016, ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε. Γι' αυτό ευχαριστούμε τους ευρωβουλευτές εκείνους που συνέταξαν τη γνωμοδότηση. Διότι την έκθεση μάλλον διορθώνει ομιλήτρια, διότι θεωρούμε ότι πραγματικά θα μας βοηθήσει. Θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις μας για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε μετά το 2016. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Εδώ θα σταματήσω. Είμαστε διάθεσή σας. Υπάρχουν διάφοροι εμπειρογνώμονες που έχουν υποβάλει κάποιες εργασίες τους. Ένα έγγραφο επαϊόντων αναφέρεται στο πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένε επιλογέ στη διάθεσή τη στην περίπτωση τη μη συμμορφώσεω. Μεταξύ άλλων ανακριβιών ε, στην έκθεση των υπερογνωμόνων... Να πω ως εκπρόσωπος Επιτροπή Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σπάνιο παράδειγμα φορέων που είναι σε θέση να, να επιβάλλουν ε, τη συμμόρφωση νομικός πώ. Και γι' αυτό και εσείς άλλωστε επεξεργάζεστε αυτό το έγγραφο. Μπορούμε νομικώ να διώξουμε του παραβάτε. Και αν είναι περιορισμένη αυτή η επιλογή κατά παράβαση διαδικασία, αν το θεωρείτε κάτι περιορισμένο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου ένα τη συνθήκη. Να εξασφαλίζουμε ότι η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και η συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, καθώ και τα μέτρα που υθετούνται δυνάμει αυτών, εφαρμόζονται ορθώ. Κάνουμε τη δουλειά μα. Και έχουμε πολύ δυνατά εργαλεία στα χέρια μα για να το πετύχουμε. Είμαστε πρόθυμοι να σα δώσουμε για άλλη πληροφορία επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Για μια ακόμη φορά σα ευχαριστώ και είναι ευπρόσδεκτη έκθεση. Ε, ευχαριστώ. Όπως πάντα λοιπόν, σε σχέση με τη συμμετοχή στι εργασίες μας, ε, για, για να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε εσεί να λάβετε το λόγο κυρία Μπέρντερ και μετά θα δούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση που είχαμε ήταν πολύ χρήσιμη και τις παρεμβάσεις ε, που ακούσαμε και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία που θα ήθελα να αναφέρω, πολύ λίγα. Σαφές όπως η κυρία Κοράτσα Μπίρτζε τόνισε, οι επιπτώσεις της μετανάστευσης ε, δημιουργεί μεταξύ των αποτελεσμάτων ευάλωτα άτομα τα οποία είναι στόχοι των ανθρωποεμπόρων και ιδιαίτερα χωρίς μικρόφωνο τώρα. Μικρόφωνο λοιπόν. Και ο αριθμός των παιδιών που αναφέρεται ότι είναι ασυνόδευτα και κινούνται ή τα διακινούν μέσα από όλη την Ευρώπη το θέμα της, ε, του εντοπισμού και ταυτοποίησης αν κάποιος μπορεί να βρει κάποια εύκολη λύση ή μια δυνατότητα καλό θα είναι, αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης με φυλάδια που καταδεικνύει ότι σε κάθε κοινότητα υπάρχει το φαινόμενο της ανθρωποεμπορίας. Υπήρχε λοιπόν ένα θύμα το οποίο επί χρόνια το κρατούσαν σε οικιακή δουλεία, σκλαβιά και το είδαμε στην τηλεόραση αυτό εδώ υπάρχουν λοιπόν εκπομπές και ειδήσει ε, σε σχέση με άτομα τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, ή δουλείας και έτσι λοιπόν μπορούν να βοηθηθούν. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και να βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα, με τους αστυνομικούς, τις διοκτικές αρχές, ε, όλους τους πολίτες της κοινωνίας που πρέπει να συμμετάσχουν για να βοηθήσουν τα θύματα να αναζητήσουν βοήθεια αλλά και να βοηθήσουν τον πληθυσμό, τους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν, να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του προβλήματος και η ανάκτηση και η επιστροφή ή η διάσωση και ε, των ατόμων αυτών πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η ε, ανάκτηση και η επιστροφή τους εκεί όπου έγιναν, αποτέλεσαν αντικείμενο ακριβώς αυτής της θυματοποίησης δεν είναι εύκολη δουλειά. Πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία να δράσουμε σε αυτό το σκέλος. Δεν είμαι ικανοποιημένη με το ποσοστό και το βαθμό υλοποίησης και εφαρμογή στην Ευρώπη σήμερα. Είναι εμβαλωματικό το έργο και αποσπασματικό και εδώ σε σχέση με την υλοποίηση που βλέπουμε ε, από πλευράς των κρατών μελών του νομοθετικού πλαισίου δεν είναι ικανοποιητική. Πρέπει τα κράτη-μέλη να καταστούν υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση και να ζητηθούν ευθύνε. Και είναι ικανοποιητικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να το κάνει αυτό για να λογοδοτήσουν και για την δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ε, επί παντός του επιστητού όπως ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική ενεργειακή εσωτερική αγορά και άλλε. Και όμως υπάρχει μια ανθούσα ε, αγορά ανθρωποεμπόρων και για το ανθρωποεμπόριο χωρίς όρια γλωσσών, συνόρων, μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους εσωτερικά στην Ευρώπη από χώρα σε χώρα, τους εισάγουν στην Ευρώπη και τους εκμεταλλεύονται. Τεράστια ποσά είναι το αποτέλεσμα αυτής της εκμετάλλευσης, ασύλληπτα ποσά. Και πώς πρέπει να δράσουμε και γιατί λοιπόν η ε, διοκτικές αρχές δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν και να ε, ζητήσουν τις ευθύνες ε, και να λογοδοτήσουν και να ε, υποστούν τις διώξεις. Πρέπει να υποστούν αυτή την ποινικοποίηση και εγκληματοποίηση και χρειάζεται αυτή η δράση από τις διοκτικές αρχές και τις υπηρεσίες διώξεως του εγκλήματος για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σίγουρα λοιπόν με πολλές παρεμβάσεις και προτάσεις ε, μπορούμε να έχουμε την υποστήριξη για να έχουμε ένα καλό, χρήσιμο, βελτιωμένο αποτελεσματικό έγγραφο στο τέλος τέλος. Και έτσι λοιπόν να πάρει αυτό στις κυβερνήσεις ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά με το σωστότερο τρόπο. Η νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπέρντερ. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Η κυρία Μπέρντερ ανέφερε το θέμα της υλοποίησης, της εφαρμογής ε, αυτής της νομοθεσίας και νομολογίας από πλευρά των κρατών μελών και ως προς αυτό περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα, στο επόμενο σημείο που είναι η παρουσίαση από πλευράς επαϊών των πραγματογνωμόνων μιας μελέτης γύρω από το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση σε σχέση με διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα, δηλαδή το εμπόριο ανθρώπων Ζητώ λοιπόν από τις ε, πραγματογνώμονες που θα κάνουν αυτή την παρουσίαση να είναι αυστηρές με τη χρήση του χρόνου από πλευρά τους. Πρέπει να τηρήσουμε τα χρονικά όρια και γι' αυτό κάθε μία θα έχει 8 λεπτά χρόνο παρέμβασης από πλευρά της. Δίνω τον λόγο στην κυρία Βάντερ Σπούλ που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ομάδας Επαϊόντων για την καταπολέμηση του ανθρωποεμπορίου από το 2003 στο 2011 έχει εξειδικευθεί στο θέμα και θα παρουσιάσει τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την κατάσταση στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Παρακαλώ έχετε τον λόγο κυρία. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή εκ μέρους της ε, καθηγήτριας που κάθεται δίπλα μου, της η οποία μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας στην έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011 από την προοπτική της διάσταση του φύλου. Υποβάλαμε την πρώτη μας ε, έκθεση ειδικά εξετάζοντας τη Γερμανία, τη Λιθανία και την Σουηδία και πιο ε, γενικά θέματα που αφορούν την οδηγία αυτή. Υποβάλαμε τη δεύτερη έκθεση για την Ολλανδία, τη Ρουμανία και το Ενωμένο Βασίλειο. Και τα γενικά μας ευρήματα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης της ε, εφαρμογής όσον αφορά την οδηγία αυτή στο επίπεδο των χωρών μελών και δεν υπάρχει συνοχή όσον αφορά τη χρήση των όρων του όρου του φίλου, αλλά καθώς και του όρου ζήτηση και θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα για τα δύο αυτά ευρήματα και η κυρία Σιβάκοβα θα συνεχίσει. Καταρχήν η χρήση της έννοιας του φίλου και την έλλειψη συνεχής όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες μέλη. Χάρη στα βρήματά μας κατά την ανάλυση ε, δομών συνδρομή στη Γερμανία, τη Λιθουανία και τη Σουηδία ε, απευθύνουμε τη σύσταση να αναθεωρηθούν οι διαδικασίε ταυτοποίηση. Ενώ η οδηγία υποχρεώνει στο άρθρο 11.2 τις χώρες μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα θύματα τη χάνουν συνδρομής αυτή τη στιγμή οι αρμόδιες αρχές έχουν επαρκή στοιχεία να πιστέψουν ότι το θύμα αυτό έχει γίνει θύμα αξιόπινης ενέργειας. Και βεβαίως η πραγματικότητα της λεγόμενης πίσιμης ε, ταυτοποίησης εντός εισαγωγικών είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική. Και πολύ συχνά ένα θύμα ε, δεν είναι εύκολο να ε, εισέλθει στις δομές συνδρομής. Αν λάβουμε υπόψη τις πρακτικές που έφερε στο φως ο φεμινισμός στις χώρες μέλη σε σχέση με τα φαινόμενα βίας κατά των ε, γυναικών. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα όσα λέχθησαν ότι ε, η εμπορία ανθρώπων είναι στο κομμάτι της δομικής βίας κατά των γυναικών. Ε, ο φεμινισμός οδήγησε πολλές χώρες μέλη να αποκριθούν να δράσουν κατά των φαινομένων βίας κατά της γυναικών γιατί πολύ συχνά υπάρχει πολύ χαμηλό κατόφλι στην ε, ενοχή κατά των φαινομένων αυτών βίας. Πολύ συχνά τα θύματα δεν αναφέρουν τις εμπειρίες τους λόγω στιγματοποίησης ή ντροπή. Γι' αυτό τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολλές χώρες ε, δεν ε, τη χάνουν ε, δεν καλύπτουν το επίσημο καθεστώς τους ώστε να τους χορηγηθεί ε, προστασία. Και αυτό έχει δυσμενεί σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στο δικαίωμα στην ε, ιδιωτικότητα και στην επιστημικότητα των στοιχείων αλλά και στην προθυμία να αποτανθούν σε αυτές τις δομές και να ταυτοποιηθούν ως θύματα σεξουαλικής βίας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ζήτησης, του όρου ζήτηση, δεν υπάρχει συνεπής ε, χρήση της σχετικής ορολογίας που να διευκρινίζεται στην λόγο οδηγίες όσον αφορά όλες τις μορφές εκμετάλλευσης που αναφέρει το άρθρο 18. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη ζήτηση ε, για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ορισμένε χώρες ε, συζητούν την ε, εισαγωγή της χρήσης των υπηρεσιών ε, ως ε, στοιχείο αξιόπινο όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία ενώ σε άλλες χώρες μέλη ορίζουν κάθε χρήση υπηρεσιών πορνείας ως αξιόπινο στοιχείο όπως γίνεται στην Σουηδία. Στη Γερμανία αυτό γίνεται υπό ορισμένε ε, προποθέσει, υπό ορισμένου όρου. Μεταξύ των που υπάρχουν διάφορε δραστηριότητε που συνιστούν ε, τη ζήτηση. Άλλες μορφές εκπετάλευσης πλην της σεξουαλικής και ζήτηση εδώ έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις στο θέμα του φύλου. Για παράδειγμα, η οικιακή εργασία όπου υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο γυναικών εργαζομένων. Και επιπρόσθετα εδώ πρόκειται για έναν τομέα όπου υπάρχει όλο και περισσότερη ζήτηση ε, φτηνή εργατική δύναμη λόγω των δημογραφικών μεταβολών σε πολλέ ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Και δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στο γεγονό της, ε, στην δυνατότητα αποθάρρυνσης τη ζήτηση σε αυτού του οικονομικού τομεί, όπω είναι ε, και εκεί βοηθεί ή σε άλλους τομείς ε, βιομηχανικούς όπως είναι για παράδειγμα επεξεργασία τροφίμων, ε, γεωργία κλπ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζιβάνκοβα για να συνεχίσει την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκριβάνκοβα λοιπόν θα λέει τον λόγο. Σίγουρα πρόφερα πολύ άσχημα το όνομά σας, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, λυπάμαι. Και για την μελέτη αυτή που θα παρουσιάσετε, θα μιλήσετε για το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν με πληροφόρησαν σωστά. Εντάξει. Thank ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Για να αποσαφηνίσουμε κάτι, όπως προαναφέρθηκε, ότι πρόσφατα κατατέθηκε για την Σουηδία, Λιθουανία και Γερμανία η μελέτη και βρισκόμαστε υπό εξέλιξη τώρα στη μελέτη, υπό ε, επεξεργασία της μελέτης για την Ρουμανία και υπόλοιπα κράτη. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, σε σχέση με το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ευρωβουλευτές μέλη της δικής σας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών γνωρίζουν το θέμα της εφαρμογής οδηγίας όπως τονίστηκε έχουν ήδη έρθει σε επαφή με αυτό. Είναι όμως θέμα των κρατών μελών να αποφασίσουν το τι θα κάνουν και βρήκαμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στην υλοποίηση αλλά και αβεβαιότητα και ανασφάλεια και περιορισμένη εφαρμογή όπως αναφέρθηκε από την κυρία Μπίρντερ ενώ οι άμεσες απαιτήσει συσχετίζουν με θέματα τα οποία δεν έχουν σαφώς καθοριστεί και επί των οποίων δεν υπάρχει κοινή συμφωνία όσον αφορά το φύλλο και τη ζήτηση όσον αφορά την ανθρωποεμπορία βρήκαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγε κατευθυντήριε γραμμές ή προσανατολισμοί για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη τη διάσταση του φύλου. Και αυτό φυσικά δυσχεραίνει την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην ε, καταπολέμηση της ανθρωποεμπορίας, δυσχεραίνει γενικά το γενικότερο πλαίσιο. Είδαμε λοιπόν ότι σε ένα φάσμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται στις γυναίκες και στα κορίτσια για θέματα πορνείας, ε, ίσως ε, είναι ένα θέμα φυσικό το ότι επικεντρώνονται σε σχέση με το εμπόριο γυναικών ε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και 2000. Τώρα όμως έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα και μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερες πτυχές και όπως επισημαίνεται στα στατιστικά της Ευρωστάτ που επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν ένα συντριπτικό στοιχείο ποσοστό για την σεξουαλική εκμετάλλευση όμως υπό την επιφύλαξη ότι είναι μια στιγμιαία απεικόνηση αυτή μια ας το πω έτσι απεικόνηση συγκεκριμένη απεικόνηση για το τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τα παιδιά. Πρέπει εδώ να μπορέσουμε να επεκταθούμε σε άλλες πτυχές για να ταυτοποιήσουμε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης που, εκμε... που ξεπερνούν την εκμετάλλευση και σε αριθμούς κιόλας του φαινομένου της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα για το 2011-2012 από πλευράς ε, ε αναφοράς ε, αριθμού μεγαλύτερου θυμάτων σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το ίδιο συμβαίνει εδώ και χρόνια κιόλα. Και πρέπει να δούμε εδώ τον επιμερισμό και την κατανομή και η πλειοψηφία μπορεί να είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, ωστόσο υπάρχει και οικιακή εργασία και η εργασία περίθαλψης και οικιακής μέρημνας που είναι δουλειά γυναικών και κοριτσιών. Θυματοποιούνται και οι γυναίκες και τα κορίτσια σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Μια από τις συστάσεις που κάνουμε στην έκθεσή μας είναι ότι η ένταξη της, ε, απαιτείται από την οδηγία πρέπει να κάνει αυτά τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές και να έχουν όλα τα θύματα ίση προσπελασιμότητα, ίδια πρόσβαση σε προστασία και υπηρεσίες όπως απαιτείται από την οδηγία. Στην έκθεση επικεντρωθήκαμε σε ένα τομέα, ένα τμήμα της οδηγίας, παροχή αρρωγής ε, και πρόληψη. Και θα πρέπει να δούμε στο σύνολο όλες τις πτυχές εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Και ιδιαίτερα επειδή μια γυναίκα, ένα παιδί, ένα αγόρι, ένα κορίτσι είναι εξειδικευμένος στόχος των ανθρωποεμπόρων για τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα άτομα αυτά ξεχωριστά το καθένα ανάλογα με τις ίδιο, ε, τα ξεχωριστά του χαρακτηριστικά και πρέπει να δούμε και τη ζήτηση φυσικά από την άλλη πλευρά. Εδώ δεν είναι χωρίς να είναι επίμαχα αυτά τα θέματα στη συζήτηση που διεξάγεται. Ωστόσο όμως σε σχέση με τους ορισμούς ε, για την ε, αναζήτηση της αλήθειας για το τι συμβαίνει και για τη μελέτη που δόθηκε υπό, σύνταξη για και την ελπίδα θα υπήρχε αποσαφήνιση για τους ορισμούς και την προσέγγιση και μια κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεισφέρουμε κατά κάποιο έστω και ίσονο σημασία τρόπο για να γίνουν πιο κατανοητά και σαφέστερα αυτά τα πράγματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σαφές στην οδηγία και η συντονίστρια της Επιτροπής για την καταπολέμηση του ανθρωποεμπορίου είπε ότι η ζήτηση υπηρεσιών κάθε μορφής και κάθε φύσης που είναι εκείνη που θυματοποιεί αυτά τα άτομα πρέπει να μας κάνει να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση αυτή σε όλες τις πτυχές ε, συλλήβδη, συνολικά καθώς επίσης και τους όρους και προϋποθέσεις που αναγκάζουν ε, τα θύματα να ε, κινούνται με αυτόν τον τρόπο και να αποτελούν μετά στόχο και να γίνονται θύματα ακριβώς και να βρούμε τις διάφορες διαστρωματώσεις από πλευράς δράσεων διότι μάθαμε ότι οι γυναίκες ε, και παιδιά που προέρχονται ίσως από το ίδιο κοινωνικό ιστό της ε, φτώχειας ε, βρίσκονται σε μια χώρα ως ε, ευάλωτη στόχη ενώ σε άλλη ίσως όχι και πρέπει να κατανοήσουμε το γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πολλές φορές εδώ χρειάζεται και ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση που πρέπει από πολλούς εμπλεκόμενους να προαθεί και μέσω των πολιτών και των συνδικών ε, και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς ε, στους οποίους ε, αποτελούν αντικείμενα εκμετάλλευσης αυτά τα άτομα και πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τι είναι εκείνο το οποίο οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έχει κέρια σημασία και σε σχέση με την Διεθνή Οργάνωση, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και σε σχέση με την περιοχή του Μεκόν στην Νοτιοανατολική Ασία και το πόσο ε, γίνονται θύματα τα άτομα αυτά. Υπάρχει το θέμα της, ε, ε, των εργαζόμενων, των πελατών που ζητούν να καταναλώσουν τέτοιες υπηρεσίες και το θέμα του ότι πρέπει να παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας σε αυτά τα άτομα και όχι να εξωθούνται σε αυτό το είδος εκμετάλλευσης ολοκληρώνω εδώ, πιέζει ο χρόνο, αλλά η έκθεσή μα είναι διαθέσιμη φυσικά σε όλου. Σα Ευχαριστώ. Eh, Σα ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Ρότ παρακαλώ. Μπεν Ρότ. Distinguished parliamentarians, ladies. Εγκεκριμένοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ σήμερα. Uh, Εργάζομαι ως σύμβουλος για τη Φινλανδία εισηγήτρια για το εμπόριο ανθρώπων. Ανεξάρτητος δημόσιος φορέας. Αρχή, στη Φιλανδία είναι αυτή. Αρκετά νομικά μέσα έχουν θεσπιστεί κατά το εμπορίο ανθρώπων. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σχετική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι ισχυρά μέσα μεγάλα επιτεύγματα. Τα θύματα ανθρωπίνου εμπορίου έχουν δικαίωμα προστασίας και βοηθείας. Να θυμηθούμε ότι κανένα άλλο νομικό πλαίσιο, όπως η καταναλιστική εργασία, η σύγχρονη σλαβιά, το πλαίσιο για τη σύγχρονη σκλαβιά, θεσπίζει τόσο ισχυρά δικαιώματα για τους ευάλωτους ανθρώπους. Η εφαρμογή αυτών των μέσων απεδείχθη προβληματική σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται τις τεράστιε διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του εκτιμούμενου αριθμού και του πραγματικού αριθμού των θυμάτων εμπορίου ανθρώπων. Και δεύτερο μεταξύ της εκτίμησης των υποθέσεων εμπορίου και τελικά των αδικημάτων που διώκονται. Ο εντοπισμό άνθρωπου εμπορίου είναι κρίσιμο σημασία. Χωρίς σωστό εντοπισμό τελικά χάνουμε στι προσπάθειε που καταβάλουμε. Τα θύματα που δεν καταγράφονται και είναι χαμηλά σε αριθμό αυτά που καταγράφονται, δημιουργούν την εντύπωση ότι το φαινόμενο είναι μικρότερη κλίμακα από ό,τι στην πραγματικότητα και έτσι δεν δίνεται σε σημασία. Τώρα, για το άτομο. Τεράστια σημασία η γυναίκα θύμα να εντοπιστεί σαν θύμα εμπορίου ανθρώπου. Διότι τότε θα έχει δικαίωμα σε βοήθεια και προστασία. Κάτι που προβλέπεται την ομοθεσία τη χώρα. Κυρίε και κύριοι. Το πλαίσιο καταπολεμήσεω του φαινομένου είναι ότι καλύτερο έχουμε στη διάθεσή μα. Υπέχουμε ευθύνη να λειτουργήσει. Πολλέ ζωέ εξαρτώνται από αυτό. Το έγγραφο αυτό που συνέγραψα και σα έστειλα αναφέρεται στου λόγου του οποίου το εμπόριο ανθρώπων που σχετίζεται με την σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί και να καταπολεμηθεί. Γενικό στόχο του εγγράφου είναι να εντοπίσουμε τα εμπόδια, συνεπώ να τα ξεπεράσουμε. Το έγγραφο επικεντρώνεται στη Φιλανδία, αλλά πιστεύω ότι πολλά από τα απορίσματα μπορούν να ισχύσουν και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η τεράστια πλειοψηφία των θυμάτων που είναι αποτελέσματα οικονομικής και σεξουαλικής εκμεταλλεύσεως είναι γυναίκες και κορίτσια. Η ανάλυση λοιπόν Πρέπει να είναι ευαίσθητο όσον αφορά τη αίσθηση του φύλου. Εγώ λέω ότι οι αντιμετωπιζόμενε δυσκολίε για την καταπολέμηση του φαινομένου, κυρίω των θυμάτων τη σεξουαλική εκμεταλλεύσεω, μπορεί να εξηγηθεί ω εξή. Πρώτον, ο ορισμό του, ανθρωπίνου, του εμπορίου ανθρώπων έχει και περίπλοκη σχέση και με την πορνεία. Και το σύστημα ποινική δικαιοσύνη δεν μπορεί να, να εντοπίσει τι ψυχολογικέ διαστάσει εκμετάλλευση και τη δυναμική τη ψυχολογική. Δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε επί το ρυσμού του εμπορίου ανθρώπων. Όταν διαπραγματευόμαστε το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για το ανθρώπινο εμπόριο, το πρώτο διεθνέ νομικό μέσο που καταπολεμά το φαινόμενο. Οι πιο σοβαρέ διαφωνίε αφορούσαν τη σχέση μεταξύ ανθρωποεμπορίου και πορνεία. Ο ορισμό του πρωτοκόλλου είναι συμβιβασμό. Συγκεράζει διάφορε απόψει περί πορνείας. Όταν αξιολογηθεί νομικά ορισμό, δεν έχει συγκεκριμένη θέση όσον αφορά την πορνεία. Καλύπτει όμως πέρα από την κατακαστική πορνεία μέσω βίας και την κάλυψη και πιο υπείων μέσων, κατάχρηση εξουσίας και ευάλωτη θέση του θύματος. Κυρίες και κύριοι, αξιοσημείωτο επίτευγμα αυτό. Πρέπει να το τονίσουμε όπως το αρμόζει. Ο ορισμός καθορίζει το πεδίο εφαρμογή. Ποια άτομα προστατεύονται και ποια χρήζουν βοηθείας. Όμως, ο ορισμός μπορεί να ερμηνευτεί τρόπο. Το πότε συμβαίνει η εκμετάλλευση και οδηγεί σε πορνεία ή άλλες μορφές εμπορικού σεξ είναι τέτοια φύσεως που δημιουργούνται αμφιβολίες κατά πόσο υπάρχει σεξουαλική εκμετάλλευση στα θύματα ανθρωποεμπορίου. Κυρίως όταν, όταν ο εγκληματίας χρησιμοποιεί ψυχολογική βία κατά των θυμάτων. Ο ορισμός του ανθρωποεμπορίου δεν χρησιμοποιείται σωστά και πλήρως. Άρα πολλά θύματα δεν εντοπίζονται ποτέ και δεν δέχονται ποτέ τη βοήθεια. Και πολλοί από αυτούς που διαπράττουν το έγκλημα ποτέ δεν προσάγονται στη δικαιοσύνη. Το σύστημα το ποινικό φαίνεται να μην εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει την όλη δυναμική της εκμετάλλευσης και τα ψυχολογικά μέσα της διάπραξης του αδικήματος του εμπορίου ανθρώπων. Αναφέρθηκε αυτό και από το Eurojust και άλλους. Εγώ λέω ότι το ανθρωποεμπόριο σπάνια είναι θέμα στιγμίας συναλλαγής, αλλά μια διαδικασία εκμετάλλευσης και υποχώρησης και παράδοσης. Το θύμα τελικά παρετείται από την αυτοδιάθεσή του, την ακεραιότητα του σώματος και την ακεραιότητα μέσω χειραγώγησης και τελικά το θύμα υποκύπτει ε, στη βούληση του θύπτη. Ανακαλύψαμε λοιπόν τα θύματα είναι από τον έλεγχο εκεί που διαπράττουν τα δίκημα παρά τα φαινόμενα φαίνεται να ζουν κανονικά, λένε θύματα. Και τα θύματα δεν έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν την εκμετάλλευση, ούτε να προστατευτούν, ούτε να ζητήσουν βοήθεια. Λόγω χειραγώγησης και ταπείνωσης που ασκεί ο εγκληματίας. Οι ειδικοί για, στην ψυχολογία και στα ψυχικά τραύματα που αναφέρονται στην εκμετάλλευση το εξήγησαν αυτό. διάφορα ψυχολογικά φαινόμενα συμβαίνουν όπως και μοιάζει αυτό το συνέστημα όπως και η διαπροσωπική βία με τον ε, σύντροφο. Πρέπει να δώσουμε προσοχή, εντοπίσουμε τα θύματα βλέποντας τις ψυχολογικές διαστάσεις του ανθρωποεμπορίου. Να καλύπτεται και στην πράξη και στην νομοθεσία αυτό. Τα στοιχεία για το ανθρωποεμπόριο τελικά βρίσκονται στα μυαλά των θυμάτων. Ε, τώρα και η, η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι δύσκολο αντιμετωπιστεί νομικά. Οι γυναίκε στο εμπορικό σεξ στην πορνεία πάντα θεωρούνται απειλέ για την κοινωνία. Η πορνεία παραδοσιακά θεωρείται σαν πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο την κοινωνία και διάφορα άλλα συμβαίνοντα όπω είναι το ήθο, δημόσια υγεία, δημόσια τάξη και ασφάλεια. Στη σύγχρονη νομική ιστορία η πορνεία οδήγησε σε νομικές απαντήσεις. Προσπαθούν να ελέγξουν τις γυναίκες πόρνες αντί να τις προστατεύσουν από την κατάχρηση και τη βία ή να καλύψουν τη ζήτηση. Αυτό τουλάχιστον συνέβη στη Φιλανδία. Το πλαίσιο για την καταπολέμηση του ανθρωποειρίου έχει ένα στόχο, να αλλάξει την όλη νοοτροπία. Θεσπίζει μέτρα βοηθείας για τους πιο ευάλωτους. Αυτό είναι μοναδικό σε σχέση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το πλαίσιο αυτό δίνει περισσότερα δικαιώματα στα θύματα σοβαρών εγκλημάτων. Περισσότερο από άλλο νομικό πλαίσιο, όπως καταναγκαστική εργασία ή δουλεία. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Η... Περιθωριοποιείται η βοήθεια προς το θύμα. Μηχανικά παρέχεται στα πλαίσια του ποινικού συστήματος και μέσω της εθνικής νομοθεσίας και στην πράξη. Τι θέλω να πω. Ότι η βοηθεία και προστασία του θύματο εξαρτάται συχνά από την ποινική διαδικασία και δυνατότητα και προθυμία του θύματο να αναφέρει αυτά που συνέβησαν σε αυτόν ή σε αυτήν και να διεκδικεί τα δικαιώματά του ή τη. Γι' αυτό πολλά τα θύματα επιλέγουν να μην εντοπιστούν, να μην ταυτοποιηθούν και δεν ζητούν προστασία ή βοήθεια. Για να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Τρίτον, σημαντικό να αναλύσουμε τι δυσκολίε που υπάρχουν αντιμετώπιση του φαινομένου σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών. Οι δυσκολίε μοιάζουν με τι δυσκολίε που έχει το νομικό σύστημα με σχέση με άλλε μορφέ σεξουαλική βία. Κυρίω αν το θύμα αρχικά είχε συμφωνήσει να συμμορφωθεί. Ακόμα και να παντρευτεί τον εγκληματία. Κυρίε και κύριοι, ελπίζω ότι αυτό το ευρύ πλαίσιο μα βοηθεί να καταλάβουμε το φαινόμενο. Γιατί ο εντοπισμό, η ταυτοποίηση του θύματο είναι τόσο δύσκολη και πώ θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Οι φεμινίστε είπαν ότι οι Φιλανδέζε που είναι ανεξάρτητες, οικονομικά ανεξάρτητες, θεωρούνται σαν υπεύθυνε και αυτόνομες και πολύ συχνά αν είναι θύματα βίας θεωρούνται ότι αυτές είναι υπεύθυνε. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στα θύματα ανθρωποεμπορίου ε, και σεξουαλικής βίας από το ποινικό σύστημα. Δηλαδή θεωρούν ότι πούλησε το θύμα σεξ Και έτσι δεν δίδεται σωστή ερμηνεία. Αν συνένεσαν μέσω τη συμμετοχή σε πορνεία οι γυναίκες δεν θεωρούνται ότι είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο ποινικό σύστημα, ανεξάρτητα αν υπήρξαν ευάλωτε και μέσα στα πλαίσια τη πορνείας και υπό ποιες συνθήκες πούλησαν σεξουαλικές υπηρεσίες. Και δεν το αναμένουμε αυτό, τέτοιου είδου ευθύνε από άλλου που είναι θύματα ε, εκμετάλλευση στον τομέα τη καταναγκαστική εργασία, Φερρυπίν. Κυρίε και κύριοι, το έγγραφο δίνει κάποιε συστάσει. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ταυτοποίηση των θυμάτων. Θέλουμε να κατανοήσουμε ότι τα θύματα ανθρωποεμπορίου έχουν δικαιώματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο χρησιμοποιώντα πολιτικά και νομικά μέσα πολιτική, ε, κοινωνική και με βάση το φύλλο. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην κατανόηση του φαινομένου και ότι παίζουν λόγο πολύ ψυχολογικοί ε, παράγοντες και μοιάζει με άλλα είδη έμφυλης βίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στοιχές. Και ποιε κοινωνικές στοιχές οδήγησαν στην αύξηση του φαινομένου και στη σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως είναι η ζήτηση για ε, σεξ με πληρωμή, αντιπληρωμής. Θέλουμε να μην είναι τόσο ευνοϊκό το περιβάλλον μέσω νομοθεσία για αυτή την πράξη. Θα πρέπει να εξολογήσουν οι χώρε τι αντίκτυπο έχουν τα μέτρα που λαμβάνουμε και αν δεν έχουμε επαρκή αποτελέσμα να τροποποιήσουμε την νομοθεσία. Τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν σε αυτό. Διότι έχει λάβει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμόσει ιδεώντα την νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πραγματικά πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας σε σχέση με τα επόμενα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η παρουσίαση, έχει το λόγο η κυρία Νούσα Τζοκόβα. Distinguished members of the... Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, έχω την ε, χαρά να σας παρουσιάσω τα προηγούμενα απορίσματα από δύο διαφορετικές ε, μελέτες στη Βουλγαρία όπου υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και οι περιφέρειες αυτές ε, αντιμετωπίζουν επίσης την εισρωή προσφύγων. Ωστόσο τα προηγούμενα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες όσον αφορά τα προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 36 ε, και στις δύο χώρες ε, ποινικοποιείται η ανθρώπινη εμπορία κάτω από τις διάφορες μορφές και στις δύο μορφές αυτές υπάρχουν, επαρκείς ε, μηχανισμοί και ε, ενεργός κοινωνία των πολιτών. Οι αρχές ε, έχουν θεωρήσει το έγκλημα της εμπορία ανθρώπων μεγάλης προτεραιότητας. Και οι γυναίκες είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των θυμάτων. Οι δύο χώρες αυτές ε, παρουσιάζουν ε, δυνατότητα προσφυγής σε ένα αποτελεσματικό ιατρικό σύστημα. Ε, υπάρχει ιατρική περίθαλψη για τα θύματα αυτά στη Βουλγαρία παρέχονται αποτελεσματικές υπηρεσίες για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και οι δύο χώρες Δίνουν προσοχή στις νέες μορφές ε, εμπορίας ανθρώπων και προωθούν την ε, έρευνα για άλλες ε, μορφές εκμετάλλευσης όπως είναι η πώληση βρεφών, η καλλιέργεια ναρκωτικών και η καταναγκαστική γάμη και όλα αυτά τα στοιχεία θα δημοσιευθούν τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια θέματα εφαρμογής τόσο σε Και αυτό, το, είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί αφορά όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όπως ανέφερα, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη Βουλγαρία. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν ε, ε κατοχυρώνονται από τον νόμο υπάρχει μια έλλειψη περικτικής ε, πολιτικής που να εγγυάται προστασία σε όλα τα θύματα. Υπάρχουν δυσκολίες να φάνε την ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αιτούντες ε, άσυλο αποκλίνονται αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει Επίσης υπάρχει έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά τις διαφορές των φύλων και έλλειψη προστασίας των δεδομένων. οι δυνατότητες συνδρομής προϋποθέτουν μια συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει επαρκής αποζημίωση προς τα θύματα, για παράδειγμα, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα στη Βουλγαρία. Υπάρχουν αφιβολίες όσον αφορά τον προσδιορισμό των ε, θυμάτων. Για παράδειγμα, example, για παράδειγμα η συγκατάθεση εκ μέρους των ε, γυναικών όσον αφορά σε ζητήματα πορνίας, όσον αφορά την ταυτοποίηση, την αναγνώριση τους ως ε, θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι αρχές λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση με τους ε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι η Βουλγαρία θεωρήθηκε ότι ε, ε, από ανεξάρτητους φορείς ότι παραβιάζει κατάφορα τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν υπάρχουν ε, επαρκείς δυνατότητες στέγασης για τα θύματα. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερων προσπαθειών επανένταξη ευάλωτων ομάδων όπως είναι η Ρωμά, κυρίως γυναικών και παιδιών υπάρχουν ζητήματα αποζίωσης, αποζημίωσης τα οποία προϋποθέτουν νέες προσεγγίσεις. Ε, παρόλο που η χρήση των υπηρεσιών σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει ποινικοποιηθεί, αυτό δεν έχει αποτρεπτική αξία. Ε, η ποινικοποίηση της ε, αγοράς ε, σεξ ε, κρίνεται ως μία αποτελεσματικό μέσο. Και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την αντιμετώπιση της πορνείας, διότι αυτό είναι το κυρίως αντικείμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να δοθεί εδώ ιδιαίτερη προσοχή. Ε, η πρώιμη νόμιμη, ε, παρέμβαση καθώς και η πρόσβαση σε νομικές ε, συμβουλές μπορούν να είναι αποτελεσματικά μέσα κατά πολέμηση των φαινομένων αυτών τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Ιρλανδία. Τα ωφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης είναι τεράστια τόσο για τα ίδια τα θύματα όσο και για τις χώρες γιατί με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μια καλύτερη πρόσβαση στα νομικά δικαιώματα των θυμάτων ε, και αυξάνονται οι δυνατότητες ε, αποζημιώσεων. Επίσης αυξάνει την πιθανότητα συνεργασίες ε, εκ μέρους των θυμάτων με τις αστυνομικές και διοκτικές αρχές. Και όταν καταχειρώνεται τα δικαιώματα των θυμάτων από τις αρμόδιες αρχές και τις διοκτικές υπηρεσίες είναι πολύ θετικότερα τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε και τους, τις τέσσερις συναδέλφους που έκαναν παρουσίαση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εργασία και εξυπηρετεί την καθημερινή μας δουλειά στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Πολύ ευχαριστούμε γι' αυτό. Για να ολοκληρώσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Η, κυρία Σακελιάδου παρακαλώ. Δύο λεπτά. Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέδρια. Σημειώνουμε με προσοχή τα σημεία που ανέφεραν οι όπως προηγούμενα σε σχέση με την συντονίστρια, σε σχέση με τις δύο παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν σε σχέση με τα κακοσκήμενα, σε σχέση με την ε, ε, νομολογία. Θα διορθώσουμε θα, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση ή σφάλμα. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε κάτι άλλο, ότι Μόνο μία μελέτη έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η μελέτη για τη διάσταση του φύλου στην, στο άνθρωπο εμπόριο που διαβιβάστηκε στην εισηγήτρια. Οποιαδήποτε άλλη μελέτη όσον αφορά γενικά τη ζήτηση δεν είναι μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ανεξάρτητες ε, πραγματονομοσύνες από διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις με βάση και υποστήριξη ευρωπαϊκή. Πρέπει αυτό να το αποσαφηνίσουμε. Έχουμε μόνο μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη γνωστοποιήθηκε και υπευλήθη στο Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο μία. Και τελευταία παρατήρηση τέλος επ' αυτού. Η ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική κατά της ανθρωποεμπορίας εντάσσει αυτό το φαινόμενο σε διάφορα άλλα όπως είναι το φαινόμενο της ασφάλειας, η στρατηγική εμπλοκή όσον αφορά την ισότητα των φύλων την πρόσφατη ε, δράση, πρόγραμμα δράσης για την δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα, πρόγραμμα δράσης, το έργο που επιτελείται για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το επιχειρήν και τις επιχειρήσεις και πολλούς άλλους τομείς που θεωρούμε ότι πρέπει να τονιστούν και να ε, συνεξεταστούν. Πιέζει ο χρόνος. Ε, Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο που μας δώσατε για να τονίσω και να πω ότι είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου ώστε να διαθέσουμε οποιαδήποτε στοιχεία όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε λέγει Πρόεδρος. Και για να ολοκληρώσουμε και πάλι προσπαθώντας να είστε σύντομοι. Κυρία Μπέρντερ έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. I Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλές πληροφορίες ε, ακούστηκαν και πολλή δουλειά λαμβάνει η χώρα. Ευπρόσδεκτο. Με ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπε η κυρία από τη Φιλανδία. Ο ορισμός της καταχρηστικής εξουσίας είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δύσκολο να βγουν, να εμφανιστούν τα θύματα γιατί ελέγχονται από τους διακινητές καμιά φορά αφαιρώντα το διαβατήριό του. Αυτό ήδη είναι αρκετά τρομοκρατικό, γιατί σου λένε μετά θα σε στείλουμε πίσω κλπ. κλπ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μια κοπέλα 13 ή 14 ετών ε, από την Ιγυρία. τη έκοψαν περίπου 2,5 εκατοστά από τα μαλλιά και τα κρατήσανε για μαύρη μαγεία. Και τη είπαν θα πεθάνει η οικογένειά σου, θα χρησιμοποιήσουν μαύρη μαγεία, θα χρησιμοποιήσουμε τα μαλλιά σου. Βλέπετε έτσι ψυχολογικά γίνονται υπόδουλοι άνθρωποι. Όταν λένε γιατί αυτά τα θύματα δεν φεύγουν και γιατί το σκάνε, ε, για αυτούς τους λόγους. Ευχαριστώ πολύ τη δουλειά που κάνατε. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Θα μπορούσα να συζητήσουμε επί ώρες. Απλώς ήθελα να τονίσω και εγώ το πόσο δύσκολο είναι τα θύματα να βγουν έξω, να αποκαλυφθούν, να αποκαλύψουν αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματο εντοπισμού και ταυτοποίηση των θυμάτων. σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπέρλε. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μια αλλαγή σε σχέση με το σημείο 11 που το 11 θα περάσει το 12 και τώρα θα συνεχίσουμε με το σημείο 12. Εδώ όσον αφορά ένα ευαίσθητο θέμα για τα ζητήματα του φίλου παρουσίαση από την κυρία Σίλβια Σουτέ όσον αφορά δηλαδή τα θέματα αυτά και μετά θα περάσουμε στη σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Σίλβια Σουτέ έχει τον λόγο παρακάτω.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 Ευχαριστώ μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και χαρά μου να παρίσταμε εδώ για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμά μου. Το αλφάβητο για ένα σύνταγμα με ευαισθησία όσον αφορά την έμφυλη διάσταση. Η φεμινιστική πρωτοβουλία της Euromed το ετοίμασε. Λοιπόν, είναι ένα δίκτυο που ζητά την ισότητα των φίλων και προωθεί τα δικαιώματα της γυναίκας στα πέσεις της δημοκρατίας. Είναι ένα δίκτυο που ενώνει στην Ευρωμοσυγειακή περιοχή διάφορες οργανώσεις. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την υποστήριξη που παρήχε μέχρι τώρα στο όλο πρόγραμμά μας ε, και από τούδε στο εξή. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα σας παρουσιάσω μια επισκόπηση. Τι κάνουμε, τι στόχους έχουμε, προς ποιους απευθυνόμεθα, ποιο είναι το περιεχόμενο, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο και ο συνάδελφος ο οποίος γκράζει θα εξηγήσει γιατί είναι τόσο σημαντικό να ολοκληρωθεί το έργο. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, στο συνταγματικό επίπεδο. Στόχος ποιος είναι. Το αλφαβήτου για το σύνταγμα που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Να, να εκπαιδεύσουμε αυτούς που διαμορφώνουν τα συντάγματα και το κοινό το πώς μπορούν να τροποποιούν το σύνταγμα, ώστε το σύνταγμα να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Να γίνονται πιο ευαίσθητα τα συντάγματα στον αφορά το φύλο. Διαφέρει είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εγχειρίδιο. Δεν είναι οδηγός για αυτού που συντάσσουν συντάγματα. Uh, Ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση. Εξετάζουμε όλε τις πτυχέ. Όχι μόνο το περιεχόμενο, την ουσία ενός συντάγματος και τη διαδικασία σύνταξης του συντάγματος και γίνεται φεμινιστική ανάλυση όλων των πτυχών. Σε ποιου απευθυνόμεθα μέσω του αλφαβηταριού του συνταγματικού αυτού. Είναι εμπειρογνώμονε. νομικοί εμπειρογνώμονε, πολιτικοί, που εμπλέκονται στη συνταγματολογία και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών και εν γέννη ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη κοινωνία των πολιτών κλπ. Να τονίσω και κάτι. Αυτές οι δύο ομάδες εκπροσωπούνται στην ομάδα που επεξεργάστηκε το αλφαβητάρι. Συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες για τα νομικά, αλλά και ειδικοί της ευρωμεσογειακής περιοχής. Κάποια μέλη είναι εδώ και στο Κροατήριο. Εκπροσωπούν χώρες όπως η Συρία, η Τινησία και άλλες χώρες της περιοχής. Απευθυνόμεθα επίσης προς τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό. Το αλφαβητάριο αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και στα διάφορα προγράμματα μαθημάτων στην ευρωμεσογειακή αυτή περιοχή, σαν εργαλείο να εκπαιδεύονται οι φοιτητέ, οι μαθητές, σχετικά με το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύνταγμα, τόσο ώστε να λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων. Να σας δώσω κάποια γεύση του περιεχομένου του αλφαβηταρίου. Περιέχει έξι κεφάλαια. Είναι απλή η γλώσσα η διατύπωση που χρησιμοποιούμε. Δίνουμε πρακτικά παραδείγματα και συμβουλές. Δίνουμε λοιπόν καλά παραδείγματα, κακά παραδείγματα. Δείχνουμε γιατί ένα σύνταγμα που λαμβάνει υπόψη στο των είναι κάτι σημαντικό σαν στόχος. Αναφέρεται στις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις των χωρών όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τη μη διάκριση που θα πρέπει αυτά να καλύπτονται τα συντάγματα τους. Αναφέρεται στις δημοκρατικές αρχές και τη σχέση μεταξύ ενός δημοκρατικού συντάγματος και ενός συντάγματος που λαμβάνει υπόψη ισότητα των φύλων. Το αλφαβητάριο αναφέρεται τη διατύπωση του συντάγματος, τη γλώσσα του συντάγματος και την ομοθεσία που απορρέει το σύνταγμα. Και δείχνει ποιε στρατηγικέ μπορούν να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί ο στόχο. Παρέχει εγγύσει για να εξασφαλίζεται ότι το συνταγματικό κείμενο δεν παραμένει κείμενο, κενό γράμμα, αλλά εφαρμόζεται. Και οδηγεί σε πρακτικές αλλαγές όσον αφορά την προστασία των γυναικών και αναφέρεται και στη δικονομία. Αναφέρεται σε όλες τις φάσεις. Μάλλον σε όλη τη διαδικασία. Πριν τη σύνταξη του συντάγματος, μετά τη σύνταξη, μετά την κύρωσή του, πώς γίνεται κινητοποίηση για τα δικαιώματα των γυναικών σε όλες τις φάσεις. Να σας πω ότι η προσέγγιση μας στην, όσον αφορά την ετοιμασία του αλφαβηταρίου ήταν πολύ πραγματιστική. Τι εννοώ. Περιμέναμε αντιστάσει. Δεν ξεκινήσαμε θεωρώντας ότι οι χρήστες του αλφαβηταρίου θα πιστεύουν ήδη στην αξία που έχει ένα σύνταγμα που λαμβάνει υπόψη την διάσταση του φύλου. Εξηγήσαμε λοιπόν γιατί είναι σημαντικά αυτά που θεωρούμε σημαντικά και τι μπορούμε να πετύχουμε εάν καταστήσουμε έμφυλα τα συντάγματα. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη πριν, που κρύβεται πίσω από το αλφαβητάρι. Ποια ήταν η μέρημνά μας. Η διαδικασία που ελπίζουμε θα ξεκινήσει η Συρία. Ετοιμασία ενός συντάγματος. Είναι ένα αλφαβητάρι που ισχύει παντού. Πρέπει να γίνει δουλειά παντού, να γίνουν έμφυλα τα συντάγματα σε όλες χώρες. Όλοι έχουμε να μάθουμε από αυτό. Τελικά, το αλφαβητάριο τονίζει ή προβάλλει τη σημασία της συνεχούς πολιτικής υποστήριξης και της πολιτικής αλληλεγγύης ούτω ώστε τα συντάγματα τα οποία συντάσσονται ή τροποποιούνται να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των ε, φίλων. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσετε κι εσείς. Α, ωραία. Μιλήστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Γυναικών η οποία μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε το αλφαβητάρι αυτό. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επί έξι σημαντικών σημείων που καταδεικνύουν το λόγο για τον οποίο πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και γιατί είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Έξι σημεία λοιπόν που συνοψίζουν το αλφαβητάρι αυτό. Πρώτον, το μήνυμα. Το περιεχόμενο του οδηγού αυτού του αλφαβηταρίου και πώς το επεξεργαστήκαμε. Το επεξεργαστήκαμε χάρη στις εργασίες ενός συμβουλίου, συμβουλευτικού συμβουλίου, που απετελείτο από εκπροσώπους τριών υπήρων, της Αφρικής, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή της Αμερικής, και είναι εμπειρογνώμονες για συνταγματολόγοι που προέρχονται από τρεις υπήρους. Η Σίλβια, αλλά και εγώ, η Σίλβια είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ είμαι από τη Συρία. Πάνω από 40 συντάγματα εξετάσαμε και μελετήσαμε. Από όλο τον κόσμο. Βλέπετε πώς η ποικιλομορφία ε, διακρίνει τις εργασίες μας. Το μήνυμα που στέλνουμε λοιπόν επικεντρώνεται επί μιας παγκόσμιας ε, αξίας, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δικαιώματα των γυναικών, και την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα αυτά ανεξάρτητα του πολιτισμού, της θρησκείας ή άλλων πτυχών. Εν ονόματι ουδεμίας θρησκείας, ουδεμίας κουλτούρας δεν θα πρέπει να υπονομεύουμε ή να παραβιάζουμε συγγνώμη τα δικαιώματα των γυναικών. Πρόκειται περί πολύ σημαντικού ε, μηνύματος στο ελφαβητάριο. Δεύτερον, χρονισμός. Η ημερομηνία που θα υποβάλουμε, θα παρουσιάσουμε το αλφαβητάριο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο σήμερα να προταθεί αυτός ο οδηγός ή αυτό το αλφαβητάριο. Πολλές χώρες και στην Ευρώπη αλλά και αλλού ε, τροποποιούν τα συντάγματά τους για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στις νέες καταστάσεις στη Συρία περνάμε μία περίοδο δυσχερέστατη. Και σήμερα είναι καλό, είναι σκόπιμο να επεξεργαστούμε ένα νέο σύνταγμα. Και σε αυτό το σύνταγμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διάσταση των φύλων. Όταν έγινε η Επανάσταση, η Αραβική Άνοιξη εδώ και κάποια χρόνια, όλος ο κόσμος ήλπιζε ότι εν λόγω Επανάσταση θα οδηγούσε σε ένα καλύτερο μέλλον για τις γυναίκες. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς λέγω, είδαμε ότι είχαμε υποχώρηση να αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και γι' αυτό είναι σημαντικό σήμερα καλό να ετοιμαστεί αυτού του είδους το αλφαβητάριο. Τρίτον, όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν τα φύλλα, Κάποιο θα πει βέβαια είμαι υπέρ της διάστασης του φύλου να λαμβάνεται υπόψη για λόγους ιδεολογικούς, θρησκευτικού, κοινωνικούς ή άλλους. Καλό αυτό, αλλά δεν πρόκειται περί γνώμης, θα πρέπει αυτά να περιλαμβάνονται στην ομοθεσία, σας συντάγματα. Εδώ, σε αυτό το αλφαβητάριο, έχουμε παρουσιάσει λεπτομερώς τις εμπειρίες από όλε τις υπήρους. Γίνεται λόγος για την σύμβαση της καταπολεμήσεως κάθε μορφής βίας και διάκρισης κατά των γυναικών ε, αναφερόμεθα εκτενώς σε αυτά, δίνουμε λεπτομέρειες στο κείμενο, αναφερόμαστε στα σχετικά κείμενα για να πούμε στις χώρες ότι πρόκειται περί υποχρεώσεως διεθνούς που υπέχουν να υπάρχει νομοθεσία η οποία σέβεται τις διάφορες αυτές προαναφερθήσεις πτυχές. Τέταρτον, μία προειδοποίηση. Πρέπει να αποφύγουμε τις παγίδες στο μέλλον. Όταν τα συντάγματα τα εξετάζουμε, μας λένε όταν καταρτίζουμε συντάγματα μας λένε να λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών, μας λένε μιλήστε μας για τα δικαιώματα των γυναικών και επικεντρωθείτε επί αυτού. Αλλά δεν μιλάμε για διαχωρισμό των εξουσιών, δεν μιλάμε για το κοσμικό κράτος, δεν μιλάμε εδώ για την κυριαρχία. Και εδώ υπάρχουν οι παγίδες. Μπορούμε να θέλουμε να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ο πρόεδρος της χώρας πρέπει να είναι άντρας. Να θα πρέπει να κηρύξει ε, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και λοιπά Να πούμε ότι στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να υπάρχουν γυναίκες. Αυτά πάντα προσέξουμε. Θέλουμε να μην υπάρχει διάκριση, να υπάρχει ελευθερία, να αποφασίζει ο λαός, να υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών, να έχουμε κοσμικά κράτη. Ε, όλα αυτά αποτελούν ε, στοιχεία που γιούνται ένα καλό σύνταγμα. Πέμπτο στοιχείο, οδηγός. Το αλφαβητάριο αυτό, οδηγός. Δεν θέλουμε να πούμε ότι το σύνταγμα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή κάλυψη, το πεδίο που καλύπτει το Σύνταγμα να είναι επαρκής. Το Σύνταγμα πρέπει να χρησιμοποιεί σωστούς όρους να επικεντρώνεται επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, να προστατεύεται η γυναίκα κατά της βίας, κατά των επιθέσεων ε, που μπορεί να υποστεί εν ονόματι θρησκειών ή κοινωνικών παραδόσεων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν φορείς που επαγρυπνούν να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα της γυναίκας. Τέλος, ο ρεαλισμός, πραγματισμός. Αυτό το αλφαβητάρι δεν ε, προτείναμε κάτι παράλογο, μη ρελιστικό, αντιθέτως. Περιγράφουμε λεπτομερώς τις εμπειρίες, τα παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να είναι υποδείγματα. Βεβαίως δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να ακολουθήσει τα υποδείγματα. Παραθέτουμε κάποια συνταγματικά κείμενα εδώ, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ε, προτείναμε κάποιες λύσεις βάσει των κειμένων, ε, και δείξαμε πως αυτά τα κείμενα θα μπορούσαν να αποτελούν εγγύηση κατά της παραβιάσεως των δικαιωμάτων των γυναικών. Αναφυσβήτητα, το απλούστερο θα ήταν να επεξεργαστούμε ε, το αλφαβητάρι. Το πιο δύσκολο είναι το μέλλον, να πείσουμε τον κόσμο να δώσει προτεραιότητα σε αυτή τη διάσταση. Μετά όταν θέλουμε να προωθήσουμε το αλφαβητάρι. Να λαμβάνετε υπόψη η διάσταση αυτή στα συντάγματα. Είμαι Σύριος, κατάγομαι από τη Δαμασκό και όταν και ξεκίνησα το εγχείρημα μου είπαν όλα αυτά τι είναι ουτοπικά και εγώ απάντησα τότε το Σύνταγμα είναι η ελπίδα μας. Ελπίδα που μας επιτρέπει να επιβιώσουμε παρά τον πόλεμο. Το Σύνταγμα είναι η ελπίδα μας μετά ε, τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Thank you so much. An enormous... Ευχαριστούμε πολύ. Τεράστια ε, συνεισφορά που μπορούμε να ε, στοχαστούμε και να προβληματιστούμε από αυτής. Ε, τεράστια πρόκληση να δημιουργηθεί ένα νέο σύνταγμα. Προέρχομαι από μια χώρα που έχει, το, ε, που έχει εντάξει και την εκκλησία, το θρήσκευμα στο Σύνταγμα και έχουμε αρκετούς ευρωβουλευτές. Η κυρία Μπιόρκ παρακαλώ, έχει τον λόγο κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ειδικά Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι που προσήλθατε εδώ απόψε. Γνωρίζω, πρέπει να πω, πόσες προσπάθειες έχετε καταβάλει για αυτό το θέμα και θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για την έμπνευση αυτή, για το μέλλον που μας προσφέρετε ώστε να υπάρξει μια προοπτική ειρήνευση μελλοντικά όταν ε, έχουμε μια τέτοια ζωφερή περίοδο που διανύουμε με την αποκατάσταση της δημοκρατίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προσπάθεια δημιουργίας μια σταθερής δημοκρατικής κοινωνίας, κοινωνίας κράτους δικαίου που θα μπορέσει να επιβιώσει και θα είναι ισχυρή και σταθερή. Είναι μια πρόσκληση και ε, πρόκληση για όλους μας ε, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε αυτό που εσείς δημιουργήσατε να το εκμεταλλευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε ώστε όλοι να μπορέσουν να συναγάγουν θετικά συμπεράσματα και να μάθουν από το έργο αυτό το δικό σας για παράδειγμα ένα σύνταγμα που θα βασίζεται και στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προοπτική ισότητα των φύλων έχει τεράστια σπουδαιότητα αυτό το θέμα. Όλα αυτά πρέπει να συναποτελέσουν τμήμα των συζητήσεων σφαιρικά που θα συνεισφέρουν και θα ενταχθούν στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις για την ειρήνευση και είναι κάτι που πρέπει όλους να μας απασχολήσει. Και μετά το έργο αυτό το οποίο επιτελείτε εσείς ε, διεξάγεται υπό τις δυσχερέστερες των συνθήκων και πρέπει αυτό να βρει μία αντανάκλαση, μία προοπτική στο δικό μας έργο να επιτευχθεί ένα καλύτερο σύνταγμα, μια καλύτερη συνταγματική προσπάθεια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στο συνταγματικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο κυρία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο υπό αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι συγκεκριμένο και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ θελκτικό και με κάνατε και ε, α, να θελήσω να μάθω και να μ, κινητοποιήσετε την περιέργειά μου. Τι γίνεται με τα 28 συντάγματα των κρατών μελών. Λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ισότητας των φύλων θα ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ώστε με αυτό το, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εξεταστούν και τα συντάγματα αυτά υπό αυτό το πρίσμα. Συγκεκριμένα δηλαδή να λάβουμε υπόψη και να δούμε τι συμβαίνει με τα δικά μας συντάγματα. Ευχαριστώ. Κάποιος, κάποια άλλη που θα ήθελε να παρέμβει. Εγώ ίσως να προσθέσω ότι ενώ συνέντασα μια έκθεση για την ΑΚΕ την κοινοβουλευτική συνέλευση ΑΚΕ και για τα θέματα των Αφρικανικών χωρών, Μαλάβη για παράδειγμα και Ρουάντα, πρόσεξα ότι υπάρχουν εδάφια και ζητούνται και για τις γυναίκες και για τα άτομα με ειδικέ ε, ικανότητες, ε, ειδικέ δεξιότητες, η ΑΜΕ ε, ποσοστώσεις. Σημαντικό αυτό σε σχέση με το έργο που επιτελούμε εδώ. Και άκουσα εκπληκτικές ιστορίες για άτομα που είναι ε, για παράδειγμα παρουσιάζονται ως ε, άτομα με ειδικέ ανάγκες και άτομα που έχουν ε, προβάλλονται ως υποψήφοι σε εκλογές. Εδώ πολλά πρέπει να γίνουν ώστε όλα αυτά για την ισότητα των φύλων να μπορέσουν να ενταχθούν, να γνωρίζει ο πληθυσμός τα σχετικά και να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ήταν και ένα από τα θέματα στο Μαλάβι όταν άτομα με ειδικέ ανάγκες δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που είχαν δικαίωμα όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Και έτσι έγινε ε, χρήση του συντάγματος ώστε να διεκδικηθεί αυτό. Είναι, έχει ρόλο ε, σημαντικό για αυτά τα θέματα μια τέτοια συνταγματική διάταξη. Αν έχει συνταχθεί με τρόπο ισοδίκαιο οι επιπτώσεις μιας τέτοιας διάταξης μπορεί να είναι τεράστιες. Είμαι βεβαία ότι ε, και στα όσα εκτέθηκαν για τη Συρία να πω ότι το ταξίδιο, η διαδρομή που θα έχετε να καλύψετε όταν θα αποκατασταθεί η ειρήνη στην ε, Συρία θα είναι τεράστια υπόθεση, θα είναι μεγάλο εγχείρημα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για την ενθάρρυνση και προτροπή σας. Τόσο πολύ χρόνο έχουμε αναλώσει εργαζόμενοι σε αυτά τα θέματα που για κάποιον που βρίσκεται εκτός όταν μας λένε ότι άξιζε τον κόπο και ήταν κάτι αξιόλογο είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Τα τελευταία δύο σχόλια το θέμα για τα συντάγματα των κρατών μελών που θέσατε ως, στην παρέμβασή σας και σε σχέση με την πρώτη παρατήρηση ναι Κοιτάξαμε, είδαμε τα συντάγματα των κρατών μελών και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο αυτό το αλφαβητάριο, αυτός ο τυφλοσούρτης πρέπει να ισχύει επί παντός ε, του επιστητού σε κάθε πεδίο. Πολλές φορές υποθέτει κανείς ότι από πλευράς συντάγματος χρησιμοποιούνται αυτά οι διατυπώσεις ως υποδείγματα για την ευαισθησία και συνειδητοποίηση του ρόλου της ισότητας των φύλων. Δεν συμβαίνει όμως αυτό και από πλευρά των κρατών μελών πρέπει να γίνει προσπάθεια. Δεν είναι ιδανικές αυτές οι διατυπώσεις και αυτά τα συντάγματα. Ίσως στην Αφρική, στην ε, Νότια Αφρική, στο Μαλάβι, στη Ρουάντα, ίσως με τη διατύπωση ε, μπορεί κανείς να καταλήξει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι γίνεται αυτό, αλλά το θέμα είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό, αυτή η θετική διατύπωση. Ίσως δεν εφαρμόζονται όλα αυτά. Λάβαμε λοιπόν όλες αυτές τις πτυχές υπόψη παρουσιάζοντας προτάσεις για αυτό το αλφαβητάριο να μάθουμε από όλες τις πλευρές πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτή τη ε, θέση ώστε το Σύνταγμα να είναι ένα θετικό μέσο και εργαλείο για να προχωρήσουμε πιο πέρα ακόμα κατανοώντας φυσικά ότι τα συντάγματα είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε για να συνεχίσουμε και λέμε στο αλφαβητάριο ότι γενικά σε ένα σύνταγμα δίνεται ολόκληρη μάχη για να συνταχθεί. Πρωτού όμως και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό τονίζουμε την εφαρμογή και υλοποίηση των νομοθετικών διατάξεων στο νομοθετικό πλαίσιο. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εγγυήσει, εχέγγυα για την εφαρμογή αυτών όλων και των αρχών που κατοχυρώνονται από ένα σύνταγμα. Ο συνάδελφος θα λάβει τον λόγο να συνεχίσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την... Ευχαριστούμε πολύ για την σας Βεβαίως ε, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις προκλήσεις. Η πρώτη είναι η διάδοση αυτού του αλφαβηταρίου, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο όρος δικαιώματα των γυναικών, η διάσταση του φύλου είναι ανύπαρκτα και δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους φορείς λήψεων αποφάσεων σχετικά με αυτή την αναγκαιότητα. Δεύτερον, η έγκριση αυτού του αλφαβηταρίου από, τους, ε, από όσους καταρτίζουν το Σύνταγμα. Τρίτον, η εφαρμογή αυτού του αλφαβηταρίου, γιατί ε, πολλές φορές είναι εύκολο να καταρτιστεί ένας νόμος, αλλά είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή του. Εμείς δεν έχουμε άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά μόνο να καταρτήσουμε αυτό το σύνταγμα το οποίο θα πρέπει να εδραιώνεται σε καθολικές αρχές και φυσικά θα πρέπει να τις σεβόμαστε. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές και στέφθηκε με επιτυχία. Ίσως ε, στη διάρκεια της δικής μας ζωής δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά, αλλά ίσως τα παιδιά μας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τέτοια συντάγματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν την διάσταση του φύλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη μελέτη για τους καταναγκαστικούς γάμους υπό το πρίσμα του φύλου και έχουμε μια παρουσίαση εκ μέρους της ε, Μαριλένα Βερμπάνη διοργανωμένη από το σωματικό τμήμα ΓΑΜΑ περιβάλλοντος. Ε, Η Μαριλένα Βερμπάνη Βερμπάρη είναι διαχειρίστρια προγράμματος και θα παρουσιάσει τα πορίσματα εν μιας έρευνας ε, την οποία ανέλαβε σε σχέση με τους καταναγκαστικούς ε, γάμους. Η Μαριαλένα ήταν επιστημονική ερευνήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο ε, για την πολιτική σχετικά με τα φύλλα στο Πανεπιστήμιο της και Επίσης ε, παρούσα είναι η κυρία Λσλέη, η οποία είναι επίσης εμπειρογνώμων και η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν λοιπόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Βερμπάνη. Ευχαριστώ πολύ. Η μελέτη αυτή έγινε μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου του 2015. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να μας δώσει μια επισκόπηση της πρακτικής των καταναγκαστικών γάμων και της ανάλυσης της ε, σχετικής νομοθεσίας στις 28 χώρες ε, μέλη υπό το πρίσμα της διάστασης του φύλου. Η καταναγκαστική γάμη αναγνωράζονται σαν μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η μελέτη εντοπίζει την έλλειψη ενός επαρκούς ορισμού των καταναγκαστικών γάμων σε ενωσιακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η συγκατάθεση για το γάμο δίνεται λόγω απειλής, βίας ή αδυναμίας λήψης απόφασης γιατί ένα από τα μέρη ε, είναι ανέλικο. Ε, η γάμη μεταξύ των παιδιών αναγνωρίζεται βεβαίως ως καταναγκαστική γάμη. Επίσης, ο καταναγκαστικός γάμος θα πρέπει να διαφοροποιείται από το γάμο που γίνεται με προξενιό. Ε, τους ε, γάμους αυτούς οι οικογένειες έχουν ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την επιλογή των ε, συζύγων. Και τέτοιου είδου γάμοι γίνονται καταναγκαστικοί όταν ασκείται κάποιος καταναγκασμός, βία ή απειλή. Ε, οι γάμοι αυτοί γίνονται... Επίσης υπάρχουν γάμοι οι οποίοι γίνονται ε, προκειμένου ε, ένα από τα δύο, ένας από τους δύο συζύγους να απολαύσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Και πάλι θεωρούνται καταναγκαστικοί όταν γίνονται υπό την ε, άσκηση βίας. Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι επηρεάζουν κυρίως τις γυναίκες. Για παράδειγμα, η το τμήμα για τους καταναγκαστικούς ε, γάμους του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι τα μεγαλύτερα ποστά αφορούν ε, γυναίκες. Ο αντίκτυπο των καταναγκαστικών γάμων ε, είναι πιο σοβαρός στις γυναίκες γιατί συχνά συμπεριλαμβάνουν σεξουαλική βία ή περιπτώσεις εγκυμοσύνης διάφορες εθνικές πρακτικές σε σχέση με τους καταναγκαστικούς γάμους υπάρχουν σε διάφορες χώρες μέλη. Ορισμένες από αυτές τις πολιτικές εφαρμόζονται στο πλαίσιο βίας ε, λόγω φύλου ή στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπινων όντων. Οι διατάξεις του αστικού νόμου διατυπώνουν ξεκάθαρες προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την κυρότητα των γάμων σε όλες τις χώρες μέλη και καθορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά την ηλικία καθώς και τη δυνατότητα παροχής ε, συνένεση στο γάμο. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διατάξεις του, του ποινικού δικαίου για τους καταναγκαστικούς γάμους στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένε ποινικέ διατάξει για του καταναγκαστικού γάμου. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων για τους καταναγκαστικούς γάμους, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει ε, μια περιορισμένη νομολογία γιατί ε, το ποινικό δίκαιο για, τα, για τους καταναγκαστικούς γάμους είναι σχετικά καινούριος σε αρκετές χώρες μέλη και πολύ σπάνια διώκονται οι περιπτώσεις καταναγκαστικού γάμου η ποινικοποίηση των καταναγκαστικών γάμων βεβαίως θα επιφέρει μακροπροθέσμως σημαντικά ωφέλη και θα έχει αποτρεπτική ισχύ για τους δράστες. Ωστόσο, η κίνδυνη αυτή ε, μπορεί να ε, προλάβουν τα, να αποτρέψουν ε, τα θύματα να αναφέρουν αυτά τα εγκλήματα και η έλλειξη δομών υποστήριξης τελικά επηρεάζει τη διαδικασία δίωξης γιατί πολύ συχνά τα θύματα δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή του ποινικού νόμου, τα οποία εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Πρόκειται για την νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τον ορισμό του καταναγκαστικού γάμου σε ορισμένες χώρες μέλη, ε, τα θύματα συχνά ε, δεν έχουν ε, τη δυνατότητα συνειδητοποίηση των έντεκων μέσων. Υπάρχει έλλειψη δομών για να υποστηριχθούν ή να συνδράμουν τα θύματα των καταναστικών γάμων και η απουσία προγραμμάτων προστασίας που να εφαρμόζονται στα θύματα των καταναστικών γάμων. Όσον αφορά τις κοινότητες των Ρωμά, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η καταναγκαστική γάμη κυρίως υπό τη μορφή ε, γάμων μεταξύ παιδιών είναι δύσκολο να ανοιχνευτεί λόγω έλλειψης ε, ε, δεδομένων για τις κοινότητες αυτές. ωστόσο η καταναγκαστική γάμη δεν είναι ένα προεξάρχον έθιμο σε όλες τις κοινότητες Ρωμά. Τώρα, όσον αφορά τι συστάσει που προκύπτουν από αυτή την έρευνα, είναι η εξή. Θα πρέπει να υιοστεί ένα κοινό ορισμό των καταναστικών γάμων σε ενωσιακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Τέτοιου είδου ορισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπω είναι ηλικία, βία, καταναγκασμό και απειλή. Οι καταναγκαστικοί γάμοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν μια μορφή βίας λόγω φύλου και μάλιστα σε όλες τις χώρες μέλη η συγκέντρωση συγκρίσιμων ε, και αξιόπιστων ε, στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθεί σε εθνικό επίπεδο. Ε, Ενδεδειγμένε υπηρεσίε υποστήριξη των θυμάτων θα πρέπει να συσταθούν ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ποινικών ε, διατάξεων να αυξηθεί και να υπάρξουν προγράμματα καταπολέμηση όλων των μορφών ε, βία κατά των γυναικών συμπεριλαμβανόμενων και των καταναγκαστικών γάμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον πολύ αυτό. Διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε διαφορετικά πολιτικά ζητήματα όσον αφορά πολιτιστικές πτυχές ε, για τις ε, κοπέλες από την Ασία που αναγκάζονται να παντρευτούν στην ε, Ινδία για παράδειγμα και σε σχέση με την αντιμετώπιση των περιορισμών για τη μετανάστευση και όλη την κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά τα κορίτσια. Θα πρέπει σε σχέση με τις οικογένειες ε, να το δούμε αυτό. Είναι δηλαδή Βρετανίδες υπήκοοι που αναγκάζονται να παντρευτούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι Ινδές υπήκοοι που θέλουν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα. Εντάξει λοιπόν, δεν έχουμε πολλούς, ε, πολλές ευρωβουλευτίνες στην αίθουσα. Έχετε κάποια σχόλια εσείς παρακαλώ. Εσείς πρώτοι. Δεν θέλω να γίνω πιεστική που ξαναζήτησα τον λόγο, αλλά θα με ενδιαφέρει συγκεκριμένα για τις, ε, τους υποχρεωτικούς γάμους αυτή η διαφοροποίηση σε, μια ένα παραδοσιακό γάμο με ή όχι ιερέα, με ή όχι τις ευλογίες της οικογένειας, κατοίκον ή όχι, αλλά σε σχέση με τον επίσημο γάμο. Μια, ένας καταναγκαστικός γάμος μπορεί να υφίσταται φυσικά, αν κάποιος ε, εξαναγκάζεται ε, να πει το ναι ενώπιον των πολιτικών αρχών ε, χωρίς να επιθυμεί να παντρευτεί όμως. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και γάμοι παιδιών που δεν μπορούν όμως επίσημα να συναυθούν. Ανεπίσημα γίνονται. Όμως η ανεπίσημη αυτή υλοποίηση ενός γάμου σε σχέση με τα παιδιά. Εκείνο που χρειάζομαι είναι πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε σχέση με αυτές τις ανεπίσημες διεξαγωγές, τελετές γάμων και το τι συμβαίνει υστερότερα όταν ακολουθεί ενδεχόμενα ένας επίσημος τυπικός γάμος είναι, ε, μετά αναγνωρίζονται επίσημα αυτές οι, αυτοί οι γάμοι. Γάμοι που έχουν ε, συναυθεί υποβία ή καταναγκασμό δεν μπορεί να επισημοποιούνται, έτσι δεν είναι. Τι γίνεται από νομικής πλευράς σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Υπό το αστικό πλαίσιο του αστικού δικαίου, οι γάμοι για τους γάμους έχουν όλα τα κράτη-μέλη διατάξεις που προβλέπουν ότι οι γάμοι θα πρέπει να συνάπτονται με αμοιβαία συνένεση και να υπάρχει ελεύθερη, ελευθέρα βουλήση η συνένεση που θα δίνεται. Σε σχέση όμως με τους γάμους παιδιών είναι άτυπη γάμοι, δεν είναι επισημοποιημένοι γάμοι, άτυπου χαρακτήρα γάμοι. Και παρουσιάζονται υπό αυτό το πρίσμα σε σχέση με τις αρχές και αυτό θέτει τις δυσκολίες διότι όταν υπάρχει εντός εισαγωγικών η συνένεση είναι δύσκολο να διερευνήσει κανείς και να διαπιστώσει αν ελεύθερα συνήφθη ο γάμος, ελευθέρα βουλήσει και συνενέσει ή όχι. Γι' αυτόν τον λόγο μία από τις συστάσεις και όρους μας προϋποθέσεις ήταν ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα θύματα τον εαυτό τους ως θύματα. Διότι αν δεν γνωστοποιήσουν στις αρχές οι οργανώσεις ε, που θα μπορούσαν να βοηθηθούν από αυτές ότι εξαναγκάστηκαν να παντρευτούν κάποιον, τι θα γίνει. Θα υπάρχει πρόβλημα να ταυτοποιηθεί και να ε, μπορέσει να αναγνωριστεί μια τέτοια περίπτωση παραβίασης των δικαίων τους, των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται λοιπόν για κέντρα όπου οι νέοι μπορούν να συνέρχονται και είναι σημαντικό αυτό να μπορούν να τοποθετηθούν έτσι. Αν επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, πρόσφατα ολοκλήρωσα μια μελέτη ολοκλήρωσα μια μελέτη στους αναγκαστικούς γάμους, για τους αναγκαστικούς γάμους στο Βέλγιο. Το θέμα του συνοικεσίου και του καταναγκαστικού γάμου τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη μελέτη είχαμε συνεντεύξεις ε, με επαγγελματίες που αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα και είπαν ουσιαστικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφοροποιήσουν μεταξύ μιας συμπεφωνημένης ε, περίπτωσης γάμου ή ενός άλλου γάμου διότι τίθεται το θέμα της ε, συνένεσης και της, ελευ... της ελεύθερης βούλησης προς συνένεση για ένα τέτοιο γάμο και του καταναγκασμού. Υπάρχει αυτή η διαφορετική τοποθέτηση ότι το συνοικέσιο, ο συμπεφωνημένος γάμος ή ο υποχρεωτικός γάμος ε, αποτελούν δύο διαφορετικά άκρα και δεν υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα να πει όχι ο υποψήφιος ή η υποψήφια που πηγαίνει να παντρευτεί υπό αυτόν τον τύπο, υπό αυτόν τον τρόπο ώστε να αρνηθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μην το δεχτεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σχέση με τον ορισμό των καταναγκαστικών γάμων αυτό και αυτό έχει ε, επιπτώσεις και στη συλλογή των στοιχείων που την επηρεάζει ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα ε, αναγκαία κατάλληλα στοιχεία για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Μετά η παιδική γάμη είναι σχεδόν πάντα, είναι πάντα καταναγκαστική γάμη. Εμπλέκονται παιδιά εδώ, ανήλικοι. Άρα λοιπόν είναι καταναγκαστική γάμη και όχι ελεύθερα βουλήση. Και ε, τρίτον, ε, η εθιμική γάμη, παραδοσιακή εθιμική γάμη. Και αυτοί είναι, θέτουν δυσκολίες, διότι γίνονται και ε, εμπλέκον, επισυμβαίνουν γύρω από έναν ιστό, κοινωνικό ιστό και παραδοσιακό πολιτισμικό ιστό. Και υπάρχει ένα καλό παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη Σουηδία αυτή η περίπτωση, όπου στην ιστοσελίδα των, α, της αστυνομίας αναφερόταν ότι ακόμα και οι εθιμικοί γάμοι πρέπει να αποτρέπονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ε, οι όσοι ε, εμπλέκονται θρησκευτικοί ηγέτες να πιστούν ότι δεν πρέπει να προβαίνουν στη σύναψη τέτοιων ε, εθιμικών ή παραδοσιακών γάμων διότι αυτοί παραβαίνουν αρχές και αξίες παραδοσιακές, ε, παραδοσιακοί τέτοιοι, τέτοιου είδους γάμοι θα πρέπει να γίνονται ενώπιον των πολιτικών αρχών και όχι μέσω αυτών των θρησκευτικών ηγετών. Μια επερώτηση, ένας γάμος που ε, αποδεδειγμένα έγινε με εξαναγκασμό αν πάει μια γυναίκα και πει ότι με εξανάγκασαν να παντρευτώ τότε αυτός ο γάμος ισχύει είναι γάμος που αναγνωρίζεται ή όχι και ακυρώνεται και μέσω αυτής της κατηγορίας και καταγγελίας ε, της εμπλεκόμενης γυναίκας που εξαναγκάστηκε να παντρευτεί ακυρώνεται θα με ενδιαφέρει να το μάθω αυτό ε αρκετές αστικές διατάξεις σε αρκετά κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν τον όρο του εξαναγκασμού ως μια προϋπόθεση ώστε να ακυρώνονται οι γάμοι, να μην αναγνωρίζονται δηλαδή ως γάμοι στη συνέχεια μέσα στα πλαίσια τα νομικά των κρατών μελών. Ναι, μπορεί να ακυρώνονται αυτοί οι γάμοι αν έχει προϋπάξει εξαναγκασμός. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θεκτικότατο, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και λυπούμε που δεν έχουμε περισσότερους ευρωβουλευτές παρόντες και ευρωβουλευτίνες παρούσες στην αίθουσα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και παρουσιάσατε το θέμα αυτό και για τον κόπο και την προσπάθεια που κάνατε. Uh, Επόμενο σημείο έκθεση της αποστολής στην Ιρλανδία. Εφτά μέλη πήγαν στο Δουβλίνο στις 24-25 Σεπτεμβρίου πέρσι. Έχετε στους φακέλους την έκθεση. Αφορά η έκθεση της επισκέψης. Αν δεν έχετε συγκεκριμένα σχόλια, δεν, θέλω, δεν βλέπω κανένα θέλει να κάνει σχόλια, άρα θεωρείται εγκεκριμένο το κείμενο σε έχει. Λοιπόν, άρα έληξε η συνεδρίασή μας. Γεια σας και καλό σας βράδυ.